Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρου των Επιτροπών προπολογισμών και Ελέγχου προπολογισμού, με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι εδώ σήμερα τον οριστέντα Επίτροπο για τον προπολογισμό και τη Δίκηση, τον κύριο Γιωάννης Χάν, σε αυτήν εδώ την ακρόαση. Θέλω επίσης να καλωσορίσω εδώ και τα μέλη της Επιτροπής Γιούρη που είναι προσκεκλημένη επιτροπή και επίσης την πρόεδρό της, την κυρία Νέθσιγκα. Υπενθυμίζω επίσης ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί τους οριστέντες επιτρόπους βάσει των γενικών του ικανοτήτων της ευρωπαϊκής τους αφοσίωσης και την προσωπική τους ανεξαρτησία. Επίσης, αξιολογεί την γνώση τους σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνουν και βέβαια και τις ικανότητες επικοινωνίας τους. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι προηγουμένω ο οριστέντα επίτροπο έχει απαντήσει γραπτά σε γραπτέ ερωτήσει που του έχουμε στείλει και οι απαντήσει αυτέ έχουν διανεμηθεί στα μέλη σε όλε τι γλώσσε. Τέλος, υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν έχει γύρει ενστάσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή ε, των ακροάσεων αυτών. Προφανώς τα επόμενα πέντε χρόνια είναι ζωτική σημασία για την Ευρώπη. Έχουμε ένα νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που πρέπει να αρχίσει να ισχύει από τα τέλη του 2020, όπω επίση και τα τομεακά προγράμματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν γρήγορα μια συμφωνία. Την οφείλουμε στους δικαιούχους και γενικότερα στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά δεν μπορούμε βέβαια να ξεχάσουμε και την ποιότητα που πρέπει να έχει μια τέτοια συμφωνία. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πιέζεται από πολλές και διάφορες πλευρές, γιατί πολλοί ζητούν ε, μείωση εξαιτία του Brexit, εξαιτία της οικονομικής κατάστασης σε εθνικό επίπεδο, εξαιτία ε, κατά κάποιο τρόπο σε τεχνητές ή παροχημένες απόψεις για ε, ισορροπημένους προπολογισμού από πλευρά των χωρών μελών και τώρα όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε για να καταλήξουμε σε πολιτικές με πραγματικά ευρωπαϊκή αξία. Θέλουμε λοιπόν μια ισχυρή κομισιόν και έναν ισχυρό επίτροπο αρμόδιο για τον προπολογισμό, χωρίς να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες μας ούτε στον ετήσιο προπολογισμό, ούτε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Περιμένουμε από τον Επίτροπο να δράσει ως πραγματικός ε, διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δρώντας μου θετερότητα και με διαβάνεια και σεβόμενο τα προνόμια και τους ρόλους του κάθε ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου, προκειμένου η συνεργασία αυτή να γίνεται μέσα σε κλίμα ε, πλήρου εμπιστοσύνη. Σίγουρα θα συζητήσουμε περισσότερο για αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια τη σημερινή συζήτηση. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Χολμάιερ για να εξηγήσει ε, εκείνη πώ θα διαμορφωθεί η σημερινή συζήτηση. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ οριστέντα πίτροπε. Τώρα, σε μένα έρχεται ο ρόλος της διάρθρωσης της συζήτηση. Ακούσαμε τι περιμένουμε ε, στο μέλλον από τον οριστέντα επίτροπο. Τώρα θα ακούσουμε τι θα γίνει σήμερα. Ο οριστής επίτροπος καλείται ε, να κάνει μια πρώτη παρουσίαση το πολύ 15 λεπτά και στη συνέχεια, στο τέλος δηλαδή τη σημερινή συνάντηση, θα έχει ακόμα στη διαθεσή του 5 λεπτά για να κλείσει αυτή την ακρόαση. Μετά την ε, αρχική του παρουσίαση θα έχουμε χρόνο για 25 ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Η συζήτηση θα γίνει σύμφωνα με το εξής ε, μοντέλο. 5 λεπτά για κάθε ε, συνολικά ερωτήσεις και απαντήσεις. Δηλαδή, ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση από τον οριστέντα επίτροπο και στη συνέχεια, αν υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση, το πολύ ένα λεπτό με ένα λεπτό μόνο για απάντηση από τον οριστέντα επίτροπο. Στην αρχή έχουμε τον πρώτο γύρο με 7 ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο δεύτερος γύρος είναι με 18 ερωτήσεις και βασίζεται στην γενική κατανομή των ερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων και εδώ συμπεριλαμβάνονται και μη εγγεγραμμένα μέλη, ενώ σεβόμαστε τον κανόνα DONT για κάθε επιμέρους κοινοβουλευτική επιτροπή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η διερμηνία σε 23 γλώσσες. Συνεπώς, όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιούν τη μητρική του γλώσσα, αλλά υπενθυμίζουμε στους ομιλητές ότι αυτά τα οποία θα πούν ε, περνάνε από διερμηνία και γι' αυτό να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα Συνήθω, όταν κάποιο ένα λεπτό προσπαθεί να βάλει δεν ξέρω πόσε ερωτήσει ό,τι έχει κάνει στο μυαλό του, μερικές φορές μιλάμε υπερβολικά γρήγορα για τους διερμηνείς μα. Οπότε σας παρακαλώ πολύ προσπαθήστε να μιλάτε με λογικό ρυθμό για να μπορούν και οι διερμηνείς να σας μεταφράζουν. Αν μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα τότε θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι στο διαδίκτυο μεταδίδονται αυτά που λέτε. Όλοι μπορούν να σας ακούσουν λοιπόν και προσπαθούν και να σας καταλάβουν συγχρόνως. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε αυτήν την ακρόαση εδώ σήμερα. Έχω εξηγήσει τα τεχνικά στοιχεία και έτσι παρακαλώ τον κύριο Χάν να πάρει το λόγο τώρα. Παρακαλώ κύριε Χάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι. Αισθάνομαι λες και γυρίζω στο σπίτι μου, θα έλεγα. Είναι μεγάλη τιμή να επιστρέφω για τρίτη φορά εδώ στο Κοινοβούλιο ως υποψήφιος επιτροπός και θυμάμαι την πρώτη μου ακρόαση, λες και ήταν χτες. Ήταν η αρχή μιας πολύ επικοδομητικής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βασισμένη σε εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό. Και αν επιβεβαιωθώ στη θέση μου, προσβλέπω στην συνέχιση της συνεργασία μας στο ίδιο πνεύμα με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερω με τις τρει επιτροπέ που είναι εδώ στην αίθουσα. Αυτή τη φορά είμαι υποψήφιο για τη θέση του Επιτρόπου για τον προπολογισμό και τη διοίκηση. Καταλαβαίνω πόσο κρίσιμη σημασία είναι να χρησιμοποιούμε του οικονομικού μα πόρου και το ταλέντο των ανθρώπων μα στο έπακρο για να ανταποκρινόμαστε στι υποσχέσει προ του πολίτε. Και είμαι δεσμευμένο να συνεχίσω να ακολουθώ το όραμα το οποίο ανέφερε στι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμέ η, πρόεδρος, η υποψήφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προκειμένου όλα αυτά να καταστούν σε αποτελέσματα, να μεταφραστούν σε αποτελέσματα. Έχουμε πολλές προκλήσει σήμερα. Οι τρέχουσε εξελίξει στην παγκοσμία σκηνή ζητούν η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο να δράσει πιο ενεργά, αλλά και να πάρει τη μοίρα στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια επιτροπή γεωπολιτική, η οποία θα ηγηθεί όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κοινωνικά κενά, αλλά και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις του αύριο, προκειμένου αυτά να καταστούν ευκαιρίες. Για μένα λοιπόν ο υπεροπολογισμό είναι μια πολιτική η οποία καθορίζεται από τους αριθμούς. Μα ε, μας δίνει δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε πολιτικέ προτεραιότητες και έτσι αποτελεί ένα από τα πιο ορατά εργαλεία για να δείξουμε στην, στους πολίτες την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προπολογισμό αποτελεί ένα εργαλείο που εξασφαλίζει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει δημοκρατικό, ε, ειρηνικό μέρος μια δύναμη ανταγωνιστικότητα και ευημερία. Είναι έκφραση τη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Παρεμβαίνει μόνο όταν είναι πιο αποτελεσματικό να δαπανηθούν χρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι στα κράτη-μέλη. Και έτσι κατοχυρώνεται στην αρχή τη επικουρικότητα και αποσκοπεί στην χορηγήση προστιθέμενης ευρωπαϊκή αξία. Αντιλαμβάνομαι ότι η επίτευξη των ε, φιλοδοξιών μα σε πολιτικό επίπεδο όπως παρουσιάστηκαν από την υποψήφια πρόεδρο εν ώψη και του Brexit και των δύσκολων διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως είπε και η Πρόεδρος, θα αποτελέσουν ένα μεγάλο ε, θέμα, μια μεγάλη πρόκληση για την ε, αποστολή μου ευθύ εξ αρχή. Ωστόσο, σας υπόσχομαι ότι δεν θα ε, εφιστούμε προσπαθειών προκειμένου να διευκολύνουμε μια επίκαιρη και έγκαιρη μάλλον συμφωνία για το δημοσιονομικό πλαίσιο και θα πρέπει να αποφύγουμε καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την εκκίνηση νέων προγραμμάτων. Μπορείτε να στηριχτείτε λοιπόν επάνω μου προκειμένου ο ο αντίκτυπο ενό προπολογισμού μικρότερο από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα υποστηρίξει ότι θα θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει αποτελέσματα. Και η, το προ, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θεωρώ ότι αποτελεί μια πολύ στεναρή βάση για συμφωνία. Η νέα πρωτοβουλία που ανακοίνωσε η υποψήφια πρόεδρο, θα πρέπει να προωθηθεί στο πλαίσιο τη συμφωνία αυτή. Αυτό σημαίνει να δώσουμε πιο συγκεκριμένη έμφαση στις ε, διαπραγματεύσεις και σε κάποια στοιχεία προκειμένου να εντοπίσουμε που χρειάζονται προσαρμοσμένες στοχευμένες προσαρμογές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σαφή θέση του που μας έδειξε ποιες είναι οι προσδοκίες σας, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Προεπιλογισμό. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Μία προτεραιότητα στις διαπραγματεύσει για το Πουδουπού θα είναι ε, το Ταμείο δίκαιη μετάβαση οι πολιτικές για να ανταποκριθούμε στην αλλαγή του κλίματος και σε αλλαγές χωρίς προηγούμενο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ενσωματωθούν η κοινωνική και η οικονομική πτυχή στην πράσινη αλλαγή από την αρχή, για να μην μείνει κανεί πίσω. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό θα καταδείξει το δρόμο και θα τροφοδοτήσει τους, ε, τα κονδύλια αυτά στι περιοχέ και στι κοινότητε που το χρειάζονται πιο πολύ. Ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό είναι ήδη ένα εργαλείο πράσινης μετάβασης. 25% των δαπανών έχει αφιερωθεί στις ε, δραστηριότητες για το κλίμα. Αύξηση κατά 25% ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό λοιπόν να εξασφαλίζει και αλληλεγγύη προς τις γειτονικέ ε, χώρες και τους εξωτερικούς ε, φορείς, ανθρωπιστική βοήθεια, διαχείριση της μετανάστευσης, αντιμετώπιση των λαθρεμπόρων ανθρώπων και άλλες πρωτοβουλίες, αλλά επίσης στρέφεται και σε επενδύσεις για το μέλλον της Ευρώπης και ε, έχω υπόψη μου την ψηφιοποίηση, την καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση. Πέρα από αυτά, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν θα πρέπει να ιδωθεί απομονωμένο άσχετα από το μέγεθο του προπολογισμού 1,1 ή 1,3 του ΑΕΠ, δεν θα αρκούσε να χρηματοδοτήσει σε καμία περίπτωση όλε τι ανάγκε και όλα τα έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό θα πρέπει να θεωρηθεί καταλήτη δημόσιων και τετικών επενδύσεων, προκειμένου να στραφούν προ τι ευρωπαϊκέ προτεραιότητες. Μόνο αν κινητοποιήσουμε όλε τι πηγέ χρηματοδότηση θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Αλλά Αλλαγή του κλίματο, καινοτομία, επενδύσει ε, και ένα κοινωνικό δίκτυο ασφαλεία. Θα ε, εξερευνήσω λοιπόν τρόπου για την καλύτερη σύνδεση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότηση, προκειμένου να πετύχουμε τι προτεραιότητέ μα και το πώ θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν η κοινή ευρωπαϊκή μας στόχη με ιδιωτικά κεφάλαια. Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά των προσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υποστηρίξουμε θα πρέπει να υποστηρίξουμε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και εδώ. Συμφωνώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι πεπισμένο ότι αν ε, συμφωνήσουμε για την πλευρά των εσόδων, θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκαθαρίσει ότι η μεταρρύθμιση των ίδιων πόρων και η διαφοροποίηση των εσόδων αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για να συμφωνήσει στο μελλοντικό πλαίσιο. Θα υπενθυμίσω λοιπόν στο Συμβούλιο τη θέση του Κοινοβουλίου και ελπίζω να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και των, του προπολογισμού με την εισαγωγή ίδιων πόρων η σωστή και χρηστή ε, χρηματοοικονομική διαχείριση και καταπολέμηση κατάχρηση πόρων θα πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, διατηρώντας την αναλογικότητα και μια σωστή, ένα σωστό επίπεδο ελέγχων. Με τον Όλαφ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε έναν ε, ισχυρό, ανεξάρτητο ε, θεματοφύλακα, ο οποίο ε, προασπίζει τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Χρειάζεται και προληπτική δράση και ισχυρή εφαρμογή σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη που έχουμε να κερδίσουμε από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Για μένα, ωστόσο, σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι ο μηχανισμός ε, κράτου δικαίου θα εξασφαλίσει την προστασία του προπολογισμού. για να ενισχύσουμε την σύνδεση μεταξύ της χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σεβασμού του κράτους δικαίου. Εδώ δεν είναι ένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων. Ο Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση. Και χαιρετίζω την, προσοχή, την ε, υποστήριξη που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση αυτή. Για τη σύγκρουση συμφερόντων θα είναι προτεραιότητά μου να παρακολουθήσω τις ε, ευρείες δράσεις τις οποίες προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2018 ο χρηματοοικονομικός κανονισμός εισήγαγε ενισχυμένους κανόνες. Θα αφιερώσω λοιπόν τους απαραίτητους πόρους για το συντονισμό των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά θέματα και υποθέσεις ε, σύγκρουση συμφερόντων και σε ό,τι αφορά την δημιουργία στενότερων σχέσεων με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε σε πρώιμο επίπεδο, σε πρώιμο στάδιο ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Ως Επίτροπος θα είμαι αρμόδιος για τη διαχείριση των εσόδων και σε ό,τι αφορά τις εισφορές των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά πειραβιάσεις στο θέμα αυτό, σε ό,τι αφορά τους ιδίους πόρους και παρακολουθεί κάθε ατασταλία. Θα συνεχίσω λοιπόν την πολιτική αυτή, προκειμένου να συνεχίσει σε καλό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να πετύχω στην ε, αποστολή μου χρειάζεται επικοδομητικός διάλογος και εμπιστοσύνη αμοιβαία. Και εγώ δεσμεύομαι για το διάλογο αυτό με τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές, με τις πολιτικές ομάδες, με μονομένους ευρωβουλευτές μέσα σε ένα ανοιχτό πνεύμα και πνεύμα εμπιστοσύνης θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε πραγματικά να αποτελέσω τον διαμεσολαβητή, τον ειλικρινή, τον αμερόληπτο μεταξύ των δύο αρχών του προϋπολογισμού. Οποιαδήποτε ανταλλαγή μεταξύ σας είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο έχω κάνει και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεσμεύομαι επίσης για να δημιουργήσω αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στις επιδόσεις των προγραμμάτων και τον δημοσιονομικό ε, σχεδιασμό την υλοποίησή τους και την υποβολή στοιχείων και εκθέσεων. Και συμφωνώ ότι ένα τέτοιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να εξαρτάται κάθε φορά από την πολιτική και να μπορούν να υπάρχουν ε, αλλαγές και διορθώσεις βάσει πάντα επιδόσεων και αξιολόγησης. Είναι πολύ βασικό επίσης αυτό που προτείνει η Επιτροπή, που είναι κανονισμό κοινών διατάξεων για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις απαιτήσει για διαφάνεια και για επικοινωνία. Εμείς έχουμε σημειώσει τις συστάσεις σας για να βελτιώσουμε την γενίκευση των εκθέσεων που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα φροντίσω να το κάνω αυτό στις ετήσιες δραστηριότητες, εκθέσεις δηλαδή κάθε χρόνο για τις δραστηριότητες της κάθε γενικής διεύθυνση και όσον αφορά τα προγράμματα και τις συνοδευτικές τους δηλώσεις στο σχέδιο προπολογισμού, όπως επίσης και ετησίως εκθέσεις επιδόσεων. Θέλουμε επίσης μία σύγχρονη και ευέλικτη δίκηση. Πράγματι, μια επιτροπή η οποία θέλει να οδηγήσει σε αποτελέσματα και να φέρει την Ευρώπη να πετύχει έναν υγιή πλανήτη σε μια ψηφιακή εποχή χρειαζόμαστε προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και γνώσεις και θα φροντίσω να γίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως θα φροντίσω να δράσω στα εξής. Πρώτον, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, καλούνται να προσλαμβάνουν προσωπικό από μια ευρεία γεωγραφική κατανομή. Σήμερα από τις χώρες που ήταν μέλη πριν από το 2004, υπάρχουν 10 χρόνια οι χώρες οι οποίες υποεκπροσωπούνται. Εγώ θα κοιτάξω να αναστρέψω αυτή την τάση. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την αξιοπιστία της δίκησης, έχει να κάνει και με την ίδια την εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεύτερον, ίσως κάτι που δεν έχει φανεί αρκετά στι γραπτέ μου απαντήσει. Εγώ δεσμεύομαι υπέρ της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων ήταν κάτι που ήταν πάντα σημαντικό για μένα. Εξυπηρετώντα τη χώρα μου ω υπουργό για την επιστήμη και την έρευνα, εγώ εισήγαγα, εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή, ε, κάποιες ε, ρήτρε με ποσοστώσεις υποχρεωτικές για τις επιτροπές και τα πανεπιστήμια. Και όταν ήμουνα στο τμήμα για την ευρωπαϊκή γειτονία, πάλι ήθελα το τμήμα μου να υπερβεί τους ε, στόχους που είχαν τεθεί. Και τρίτον, θα φροντίσω για τη διαφάνεια, την ακαιρότητα, τη λογοδοσία, τον επαγγελματισμό και την ε, δέσμευση υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αν ε, οι Ευρωπαίοι θέλουμε να έχουν και να εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να φροντίσουμε. Και αν εμπεβεβαιωθώ στη θέση μου, θα φροντίσω να βρω τον τρόπο για να έχουμε ε, προσωπικό υψηλών προδιαγραφών. Και τέταρτον, δεσμεύομαι να φέρω αποτελέσματα και όσον αφορά την ψηφιακή τροποποίηση της Κομισιόν, δηλαδή να έχουμε λύσεις στην δημόσια δίκηση που να έχουν να κάνουν με τα δεδομένα και τον ψηφιακό κόσμο. Να εξυγχρονίσουμε επίσης την υποδομή μας με έναν ασφαλή τρόπο. Θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτελεί το παράδειγμα και να συνεργάζεται με τις χώρες μέλη για να αλλάξει ο ευρωπαϊκός δημόσιος τομέας και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Τέλος, θα διασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και τις ικανότητες να πετύχει αυτή την ψηφιακή μετάβαση, χωρίς βέβαια να θέτει τον εαυτό της σε κίνδυνο. Εν κατακλείδη, προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί σα ω επίτροπο αρμόδιο για τον προπολογισμό και την Δίκηση, προκειμένου μαζί να φέρουμε αποτελέσματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμεί, βάσει των φιλόδοξων πολιτικών μας στόχων. Και τώρα περιμένω τι ερωτήσει σα και προσβλέπω επίση σε μια ενδιαφέρουσα και καρποφόρα συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Χάν και σας ευχαριστώ και για το γεγονό ότι σεβαστήκατε και το χρονικό όριο. Θα ζητήσω από όλους τους ομιλητές να κάνουν το ίδιο. Και στο πρώτο γύρο λοιπόν ερωτήσεων θα δώσω το λόγο στον κύριο Χωσέ Μανουέλ Φερνάνδες από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Και θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Καταδεικνύει την ε, εμπειρία που έχει ήδη ο υποψήφιος επίτροπος σε ό,τι αφορά τα θέματα του χαρτοφυλακίου του και πραγματικά ότι έχει μεγάλο επίπεδο φιλοδοξίας και αυτό ε, συνάδει με αυτά που έχουμε ακούσει. Τον ε, Νοέμβριο του 2018 το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια εντολή με τεράστια πλειοψηφία σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και σε ό,τι αφορά το σύστημα ιδίων πόρων. Εμείς λοιπόν από τότε είμαστε έτοιμοι και προτιθέμεθα να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Περιμένουμε ωστόσο το Συμβούλιο ακόμα. 1,3% του ΑΕΠ για 27 κράτη-μέλη. Αυτός ο αριθμός δεν είναι τυχαίος. Αυτό το 1,3% αποτελεί αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε βάσει λογικών ε, υπολογισμών. Προσθέσαμε τα ποσά που χρειάζονται για κάθε πολιτική. Έχουμε τις υφιστάμενες πολιτικές, την κοινή αγροτική πολιτική, την κοινή ελευθερική πολιτική, όλα αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν. Αλλά έχουμε και άλλε πολιτικέ οι οποίε ενισχύονται. Το εράσμο, το περιβάλλον, η έρευνα, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αν τα προσθέσουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί, καταλήγουμε στο 1,3% του ΑΕΠ των 27 κρατών μελών. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που έχω να σα κάνω είναι η εξή. Συμφωνείτε με την πρότασή μα, συμφωνείτε με τη μεθοδολογία μα εδώ στο Κοινοβούλιο. Μια μεθοδολογία bottom-up και συμφωνείτε και με την εξή δήλωση ότι νέες προτεραιότητες θα πρέπει να ακολουθούνται με νέα ε, χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Εκτός για Επιτροπός. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προηγούμενους ε, που ήταν από εμά για την ε, πολύ ρεαλιστική και καλή αυτή ε, προσέγγιση. Συμφωνώ, χρειάζεται μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, bottom up, για να δούμε τι χρειάζεται. Αλλά και ανάποδα να το πάρουμε από πάνω προς τα κάτω σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές. Ποιες είναι οι οδηγίες που μας δίδονται. Σε ένα ιδανικό κόσμο αυτά τα δύο συναντώνται σαν μια σύραγγα η οποία οικοδομείται. Ξεκινάμε από τι δύο πλευρέ και συνδυόμαστε στη μέση. Ε, πριν από 6-7 χρόνια έκανα κάτι παρόμοιο άλλωστε. Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Πολιτική συνοχή. Ακολουθώντα από κάτω προ τα πάνω την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για το 2020, αλλά ξεκινήσαμε επίσης από κάτω προς τα πάνω να επισκευάζουμε αν θέλετε, τα μεμονωμένα προγράμματα και τότε για πρώτη φορά εισήχθη για πρώτη φορά ένα ελάχιστο ποσοστό χρημάτων το οποίο θα έπρεπε να δαπανηθεί για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ο σωστό τρόπο να υπάρχει μια προσέγγιση από κάτω προ τα πάνω και μετά να δούμε πού καταλήγουμε και να προσπαθήσουμε στη συνέχεια να κάνουμε διαπραγματεύσει. Ελπίζω το μοντέλο αυτό να πείσει και τα κράτη-μέλη μας και ιδιαίτερω εκείνου που είναι πιο διστακτικοί και αποκοινούμε του συναδέλφου τους μας θα προσπαθήσουμε να πείσουμε εκείνους ιδιαίτερα που έχουν εστιαστεί στο 1% προκειμένου να δούμε τι γίνεται με τις νέες προκλήσεις που χρειάζονται πιο πολύ ευελιξία. Η συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Φερνάνδες. Θέλουμε μία συμφωνία σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά και τους ίδιους πόρους και Στηριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πείσει τα κράτη-μέλη. Ποιε είναι λοιπόν οι. Σε τι ύψο φαντάζεται του ίδιου πόρου ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι υποστηρίζετε εσεί ω Επιτροπή, όπω γνωρίζετε. Ο επίτροπο, ε, Εδώ έχουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένε ε, ιδέε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το φόρο για τι πλαστικέ σακούλες, για την επέκταση των δικαιωμάτων στα πλαίσια του προγράμματο εμπορίου Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα των εσόδων από το σύστημα ETS, λοιπόν, εδώ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ γρήγορα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουμε και κάποιους άλλους ίδιους πόρους όμως. Προς το παρόν δεν είναι ρεαλιστικό να ελπίζουμε συμφωνία επ' αυτών. Αλλά είμαι ιδιαίτερα δεσμευμένος. Ίσως να έχουμε και άλλες ευκαιρίες μέσα στην ακρόαση να το συζητήσουμε. Είμαι πολύ δεσμευμένος λοιπόν για να επεκτείνουμε τους ίδιους πόρους σε ό,τι αφορά το συνολικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εντοπίσουμε ενδεχόμενους ίδιους πόρους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι πρωτοβουλίε για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματο. Σα ευχαριστούμε πολύ. Η δεύτερη ερώτηση είναι από την κυρία Καρδιαθαβάλ Ρούμπιαλ, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Οριστέντε Επίτροπο, λέγατε ότι έχετε μεγάλη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα όμως σας ανέθεσαν την ε, λιγότερο, το λιγότερο εύκολο θέμα. Γιατί? Γιατί όλοι υπόσχονται, αλλά κανένας δεν σκέφτεται πώς θα χρηματοδοτηθούν οι υποσχέσεις αυτές που κάνουν. Εμείς έχουμε σημειώσει τις διάφορες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Μετάβασης, για το αέρασμος, τη Νεολαία κτλ. Διάφορες προτάσεις που όμως δεν είναι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρόκειται μόνο για πρόταση της νέας Προεδρού, αλλά και πολλοί υποψήφοι επίτροποι έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν με τις προτάσεις αυτές. Συνεπώς εδώ υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις συγκεκριμένες προτάσεις για τον επόμενο προπολογισμό. Συνεπώς, δεν πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να υποβάλει μια νέα πρόταση προσαρμοσμένη, ώστε να δείξει ότι εκτός από λόγια υπάρχει και συγκεκριμένη δέσμευση με νούμερα. Και στην αρχική σας παρουσίαση ακούσα το Targeted Adjustment. Όταν μιλάμε για διορθώσεις, συνήθως μιλάμε για περικοπές. Και το είπε και ο Χωσέ Μανουέλ, δεν μπορεί να έχουμε νέε προτεραιότητε με λιγότερα χρήματα. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό εφόσον επιβεβαιωθείτε στη θέση του Επιτρόπου. Απάντηση. Επαναλαμβάνω, θα έλεγα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια πολύ δυνατή βάση, η οποία ακολουθεί μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την πρότασή του και ιδανικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα σημείο διαπαφή μετά των δύο αυτών προτάσεων, προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία θα απασχολήσουν και την Μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά που έχει ορίσει και η Μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προτεραιότητε. Ένα μεγάλο τμήμα λοιπόν αυτών θα το πετύχουμε με μια προσαρμογή του υφιστάμενου προπολογισμού. Αυτό είναι εφικτό, είναι δυνατόν. Φυσικά υπό τον όρο ότι δεν θα πέσουμε σε καμία περίπτωση κατά από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτό δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα λειτουργήσει. Αφενός λοιπόν έχουμε τις ε, συζητήσεις με κάποια κράτη-μέλη, όχι με όλο το Συμβούλιο, γιατί πολλά κράτη-μέλη μας υποστηρίζουν, σαφώς σε ό,τι αφορά τα μέσα που χρειαζόμαστε. Και όπως σας είπα, ένα ταμείο δίκης μετάβασης ε, μπορεί να διαμορφωθεί με κάποιες προσαρμογές του προϋπολογισμού και το σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης. Και αυτό είναι υλοποιήσιμο. Υπάρχουν πολλοί, στομί, πολλοί τομείς, λοιπόν, τους οποίους θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε με μια ισχυρή ένα ισχυρό καθορισμό των προτεραιοτήτων. Αν είμαστε λοιπόν πολύ αυστηροί, μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες τώρα και το reporting, την υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να επιμείνουμε εκεί που είναι αυτό απαραίτητο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα μέτρα μας για την αλλαγή του κλίματος, προκειμένου όλα αυτά να υλοποιηθούν όπως έχουμε προγραμματίσει. Συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μα το πρόβλημα είναι ότι αν θέσουμε προτεραιότητες, άμα τις προσθέσουμε όλων των επιτρόπων της προτεραιότητες και όλων των χωρών μελών, συν εκείνες του Κοινοβουλίου, ε, δεν βγαίνει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για σας και καλό θα ήταν να βοηθήσετε το Κοινοβούλιο για να έχει καλά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις. Τώρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Σκέφτεστε εσείς κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία με δείκτες που να μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε κατά πόσο το δημοσιονομικό πλαίσιο όντως πετυχαίνει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά που ανέλαβε και η νέα πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, υπόσχομαι εδώ το εξή ότι θα πάω σε όλες τις πρωτεύουσε και θα δώσω προτεραιότητα στις ε, πρωτεύουσε εκείνες που ανακοίνωσαν ότι θα υποστηρίξουν ένα πολύ πιο χαμηλό επίπεδο προπολογισμού για να εξηγήσω τι ακριβώ χρειάζεται, να είμαι σε επαφή και με την κοινή γνώμη, να βρω συμμάχου. Ήθελα να κάνω και κάποιε κινήσει προ την κατεύθυνση αυτή. Βλέπουμε λοιπόν τις ε, βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την προστασία του κλίματος που είναι επιθεμητές. Θα πρέπει να διατεθούν πόροι προς την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων. Καταρχάς, ε, αυτό είναι θέμα πολιτικού σχεδιασμού. Βάσει αυτού έχουμε το πλαίσιο απόδοσης, performance framework, όπου και εδώ υπάρχουν δείκτες για τα φύλλα σε ό,τι αφορά τον τομέα της έρευνας, του εράσμους κτλ. Και το λέω ξεκάθαρα. Αν υπάρχουν εδώ ελλείψεις που θα εντοπίσουμε στην ενδιάμεση ελευθέρωση, θα πρέπει να υπάρξουν και αντίστοιχε προσαρμογέ. Ευχαριστώ. Βαλερή Χαϊέ για το Renew. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Χάν, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Θέλω να επιμείνω εδώ επί ενός θέματος πολύ σημαντικού για το Ευρωκοινοβούλιο που ήδη αναφέρθηκε. Αναφέρει τους ίδιους πόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πετάπητος ε, πολλές διεξόδους για νέους πόρους κυρίως μέσω του συστήματος ανταλλαγής ε, εκπομπών διεξοδίου του, ε, του ή για το ποστό του, του, του πλαστικού. Η κυρία Βαντελάιν υποσχέθηκε να θέσει φόρο άνθρακα στα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισπίζεται του ίδιου πόρου, του πράσινου, είναι έτοιμη από τον Νοέμβριο του 2008 για αυτά τα θέματα. Στο Συμβούλιο οι συζητήσει σε αυτό το θέμα είναι μετριοπαθεί, θα έλεγα, και δυσανάγνωστε. Υπάρχει μεγάλη αδράνεια και το Κοινοβούλιο αποφάσισε την έγκριση του επόμενου δημοσιονομικού πλαίσιου να το διασυνδέσει με τη δημιουργία νέων πόρων. Ε, κύριε Χάν, το μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο θα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα που ζητούν ακριβεί απαντήσει. Καταρχά, ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία θέτουν τροχοπέδι στην πρόοδο όσον αφορά του ιδίου πόρου που είναι πράσινοι. Και δεύτερον, ποια επιχειρήματα θα προωθήσετε για να πείσετε αυτέ τι χώρε. Και ειλικρινά, θα είσαστε σε θέση να ασκήσετε πιέσει επί του Συμβουλίου, ούτω ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το θεμελιώδε χαρτοφυλάκιο για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα και εισαγωγικά και στην απάντηση της πρώτης ερώτησης, έχουμε κάποιες προτάσεις για νέους ίδιους πόρους που έχουν εξεταστεί επεσταμένως στην πολιτική συζήτηση. Καταρχάς, ο φόρος, το τέλος για τις πλαστικές σακούλες. Εδώ υπάρχει επί της ουσίας ήδη μια συμφωνία. Νομίζω μια χώρα διστάζει η Πολωνία. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ε, το πρόβλημα αυτό θα ξεπεραστεί, φαντάζομαι. Ήδη υφίστανται δημοπρασίες για το σύστημα εμπορίας ρήπων, το ETS. Θέλουμε μεγαλύτερο ποσοστό. Και εδώ πάνε καλά οι συζητήσει. Και επίσης υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα για το πρόγραμμα αυτό εμπορίας ρήπων να επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως για παράδειγμα στον, στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, των θαλάσσιων μεταφορών και εδώ λοιπόν ε, θέλουμε ανοιχτό πνεύμα από το Συμβούλιο. Είναι διαφορετική τώρα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το CCTP. ένα τέλος για τις ε, διασυνοριακές ε, εταιρείες συναλλαγές. Εδώ υπάρχει ως επιτοπλίστων ε, διστακτικότητα από τα κρατη Και εδώ νομίζω ότι θα χρειαστεί να υποβάλουμε καινούργια πρόταση στο μέλλον. Η κυρία Φοντεν η υποψήφια πρόεδρος, ανέφερε και τον φόρο τον διασυνοριακό για τον άνθρακα. Αυτό εκ πρώτης όψεως ε, το υποδέχονται πολύ θετικά, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό στην πράξη. Για να συνοψίσω, οι πιο συγκεκριμένες ε, προτάσεις που έχουμε υπόψη μας ε, βραχυπρόθεσμα είναι το θέμα του ETS και το τέλος για τις πλαστικές σακούλες. Η διευκρινιστική ερώτηση, συμπληρωματική μάλλον. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά δεν απαντάτε στις ερωτήσεις μου, κύριε Χάν. Αναφερθήκατε στην Πολωνία. Πολύ καλά. Σίγουρα και άλλα κράτη-μέλη θέτουν τροχοπέδι στο ζήτημα. Και είναι σημαντικό να ρίξουμε το φως στο σχετισμό δυνάμεων στο θέμα αυτό. Να υπενθυμίσω ότι η συνεργογική σα ομιλία αναφερθήκατε ότι είναι αναμφισβήτητη και σταθερή η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα εγκρίνουμε το επόμενο μισονομικό πλαίσιο χωρί να υπάρχουν νέοι ίδιοι πόροι. Αν υπάρχει μπλοκάρισμα, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο επίγουσα ανάγκη για να δρομολογηθούν τα προγράμματα. Θα είναι κάτι απαραίτητο να προστατευτούν οι δικαιούχοι. Σα ρωτήσαμε γραπτό για το θέμα και η απάντησή σα δεν υπήρξε πιστική. Επίση, θέτω και το εξή ερώτημα. Μπορείτε να μα εγγυηθείτε σήμερα ότι θα παρουσιάσετε ένα τέτοιο σχέδιο για να παραταθούν τα προγράμματα και δεν σα μιλάω για το άρθρο 312 παράγραφος 4 τη Συνθήκης λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και εντό τη καλύτερη δυνατή προθεσμία, ούτως ώστε να εγκριθούν αυτά εγκαίρω και να προστατευτούν οι δικαιούχοι. Επαναλαμβάνω, για να μην υπάρξει παρανόηση. Είμαι στο πλευρό σας και παραπάνω σε ό,τι αφορά το θέμα των ίδιων πόρων, νέων ε, επιπρόσθετων ίδιων πόρων και η τρέχουσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θα εφαρμοζόταν, θα προέβλεπε το ποσοστό των ίδιων πόρων στο συνολικό προπολογισμό να πάει να αυξηθεί κατά πάνω πάνω από 25%. Έχω χρόνο, μάλιστα. Γιατί η δεύτερη ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο εξή. Από κοινού να εφαρμόσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις το contingency planning, αυτό το σχέδιο και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, θεωρώ ότι είναι η τελευταία λύση. Αν δεν καταφέρουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Εγώ προσωπικά θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και αυτό σημαίνει δηλαδή το αργότερο το χειμώνα να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα τέλη του χειμώνα. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα τώρα να αρχίσουμε να μιλάμε για σχέδιο Β με μια εναλλακτική λύση, γιατί αυτό θα αφαιρέσει την πίεση που θα έχουν οι διαπραγματεύσεις. Και αν θέλετε λοιπόν να κάνετε μια πρόταση για σχέδια έκτακτης ανάγκης, ε, κινητοποιούμε τη θεσμική κατάσταση, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δηλαδή, θα πρέπει να υποβάλουν την τοποθέτησή τους εκ νέου και αυτό θεωρώ ότι θα αποσπάσει την προσοχή από το βασικό στόχο που είναι να διαμορφώσουμε και να συμφωνήσουμε για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Και θα σήμαινε ότι όλοι οι στόχοι τους οποίους ε, θέλουμε να πετύχουμε, να κάνουμε πιο πολλά για την αλλαγή του κλίματος, για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, ότι όλα αυτά θα πάρουν ε, μία αναβολή ενός έτου. Σας παρακαλώ λοιπόν, είμαι στο πλευρό σας να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε για το πολιτισμικό πλαίσιο και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και τα μέτρα αυτά να στα για μέτρο τελευταίας διαφυγής. Εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστώ. Ράσμους Άντρεσεν για τους Περασίνους. Θα μιλήσω γερμανικά. με κύριε Χάνα, το κλίμα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και θα πρέπει να κάνουμε σαφώς πιο πολλά προκειμένου να σταματήσουμε την κρίση του κλίματος. Εμεί οι πράσινοι πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει μόνο αν διαμορφώσουμε τη διαφορετικό τρόπο τον προπολογισμό και το σύστημα χρηματοδότηση. Δεν φτάνει να παραμείνουμε στην παλιά μας πολιτική. Θα πρέπει κάτι να αλλάξει. Συγκεκριμένα λοιπόν, τι προτάσεις έχετε για να αποτυπωθεί αυτό στο πολιτισμό- πλαίσιο. Είμαστε αντιτεθειμένοι να ξεπεράσουμε και αυτό το 25% σε ό,τι αφορά τα μέτρα για το κλίμα, αν δεν αρκέσει αυτό το 25% του προπολογισμού. Και συγκεκριμένα, θα υπάρχει αξίωση να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο για τη φύση. Θα συμφωνούσατε με αυτή την πρόταση. Απάντηση. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ήδη μία πρόταση σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα να είναι στο 25% του προπολογισμού. Η αύξηση αυτή είναι κατά 25% σε σχέση με την υφιστάμενα επίπεδα. Με το υφιστάμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι φιλόδοξη η αύξηση. Έχετε δίκιο ωστόσο. Δεν θα το τέλος της διαδρομής αυτής ούτε επιτρέπεται να είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι σημαντικό λοιπόν καταρχάς να πετύχουμε αυτό το 25% στα μεμονωμένα προγράμματα. Στον τομέα των αγροτικών, για παράδειγμα, προβλέπουμε 40% των μέσων να χορηγηθεί σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος. Στο Περιφερειακό Ταμείο 30%, στο Ενέρευνα 35%, Γειτονία και Διεθνή Συνεργασία 25%, με Ταμεία σε 37%, Connecting Europe Facility 60%. Άρα προβλέπονται ήδη πάρα πολλά. Το θέμα είναι τώρα πώς στα μεμονωμένα προγράμματα, είτε μέσω άμεσης διαχείρισης θα γίνει αυτή η αύξηση, είτε σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κοινή διαχείριση να οριστούν πραγματικά αυτά τα επίπεδα. Εκεί θα επικεντρωθούν οι συζητήσει του επόμενου μήνε και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όσο πιο γρήγορα να έχουμε στα χέρια μα το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να ξέρουμε τι ισχύει σε τομεακό επίπεδο και βάσει αυτών να κάνουμε τον προγραμματισμό μας από το παρελθόν μου και την εμπειρία μου ως Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης έχω ζήσει να έχουμε μόνο 14 ημέρες μετά την λήξη των διαπραγματεύσεων και φυσικά αυτό έχει συνέπειες για την απορρόφηση των κονδυλίων. Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί αυτό για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους φιλοδοξούς στόχους μας. Και θα πρέπει οι μελλοντικέ λοιπόν συζητήσεις εκεί να επικεντρωθούν. Εγώ θα έλεγα και ζητώ αυστηρό προγραμματισμό και καθορισμό προτεραιοτήτων. Αν δεν λειτουργήσει αυτό και επικρατήσει η άποψη ότι πρέπει να γίνουν προσαρμογές, ε, θα είμαι ο πρώτος που θα το υποστηρίξει. Ευχαριστώ πολύ. Στην πληρωματική ερώτηση τώρα. Σας ευχαριστώ. Δεν απαντήσατε ακριβώς αυτό που ρώτησα, αλλά πτύφεται και το θέμα των επενδύσεων, πέρα από τις επενδύσεις μάλλον, τίθεται και το θέμα του πώς θα δαπανούνται οι πόροι και κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσαρμογή στο κλίμα. Τίθεται το θέμα και των ορεκτών ε, πόρων και των προγραμμάτων που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές επιχειρήσεις ε, βγαίνουν από ορυκτά, από επιχειρήσεις που έχουν ορυκτά καύσιμα. Και η Eurocola, το λόμπι για τον άνθρακα, λαμβάνει χρήματα από την Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Προτίθεστε λοιπόν να δώσετε μεγαλύτερη διαφοροποίηση στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, προκειμένου να μην χρηματοδοτούνται τέτοια προγράμματα. Απάντηση. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος του Ταμείου Δίκης Μετάβασης. Ε, τουλάχιστον οι περιφερειές εκείνες που έχουν ε, μεγάλη επιβάρυνση από το διοξείδιο του άνθρακα. λόγω της παραγωγής ενέργειας ε, βάσει άνθρακα, να τις βοηθήσουμε να απομακρυνθούν από την παραγωγή ενέργειας με τον τρόπο αυτό και να περάσουν σε άλλους τρόπο παραγωγής ενέργειας ή γενικώ ε, οικονομικής αξιοποίησης της περιοχής. Να διαθέσουμε λοιπόν επίσης ε, μέσα, ήδη υπάρχουν μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τραμείο σε ό,τι αφορά την ε, εναλλακτική κατάρτιση των ανθρώπων αυτών. Συχνά αυτά τα εργοστάσια βρίσκονται και σε μέρη όπου υπάρχει και έντονη δραστηριότητα ανθρακορίχων και οι ανθρακορίχοι λοιπόν θα πρέπει να επανακαταρτιστούν. Ακριβώ αυτό είναι ο στόχο του Ταμείου τη Μετάβαση. Θα στο λέω όμω ότι δεν πρόκειται να φτάσει το Ταμείο αυτό. Θέλουμε ένα ακριβή προγραμματισμό σε ό,τι αφορά τον Ταμείο Συνοχή, τα Ταμεία Καταστατικά. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, αλλά κάνουμε και συζητήσεις με τον κύριο Τίμερμαν για το θέμα αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια συνέπεια σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προωθούμε. Um, uh, για το ID. Εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και εγώ γερμανικά θα μιλήσω, κύριε Χάν. Δεν θέλω πιο πολλά χρήματα να μου δώσετε. Το αντίθετο, εμένα με πιέζει κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο με απασχολεί. Είμαι εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμού και Ελέγχου του Προπολογισμού και συχνά αντιμετωπίζουμε το εξή πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι πραγματικά λυπής και υποφέρει και αυτό φαίνεται ιδιαίτερος στην χορήγηση απαλλαγής στο άρθρο 261 κατοχυρώνεται η χορήγηση απαλλαγή αυτή. Ε, επί 9 χρόνια λοιπόν αρνείται το Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή. Ερωτώ λοιπόν το εξή. Τι θα κάνετε, τι μέτρα θα λάβετε προκειμένου αυτή η απαραίτητη συνεργασία να βελτιωθεί και προκειμένου να εξασφαλίσουμε στο μέλλον την διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Μιλάτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας χωρίς απαλλαγής. Όχι, να λάβει χώρα. Επί εννέα, χώρα, επί εννέα χρόνια το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απαλλαγή. Το Συμβούλιο. Να σας διαβάσω το άρθρο 261. Η απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά τους λογαριασμούς για όλα τα έσοδα και όλες τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση περιλαμβάνει όλα τα θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο λοιπόν θα πρέπει να λάβει απολαγή και δεν συνεργάζονται. Κοιτάξτε, με πιάνετε εξαπίνης. Πρέπει να το εξετάσω αυτό. Γιατί δεν είναι... Είναι απαράδεκτο αυτό. Εγώ διαρκώς ασχολούμαι με θέματα ε, χορηγής απαλλαγής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ θετικά, πρέπει να πω και νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο μπορούμε αμφότεροι να είμαστε περήφανοι. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, δεν θα διστάσω, γιατί είμαι υπεύθυνο για όλο το προπολογισμό. Θα κάνω λοιπόν εντατικέ συζητήσει προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Άλλη μια ερώτηση. Προηγουμένως είπατε κύριε Χάν ότι θέλετε να επιτηρήσετε το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλετε να προχωρήσετε ακολουθώντας το καλό παράδειγμα. Αυτό με απασχολεί ιδιαίτερος λοιπόν. Να το πάρετε στα σοβαρά. Να σας καλέσω και να σας ζητήσω να μου πείτε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις όπως αυτή που περιγράψαμε πριν από λίγο και δεν μπορούμε να είμαστε ο εισαγγελέα του φορολεγούμενου. Γιατί το κράτος δικαίου και η νομοθεσία την οποία εμείς περάσαμε δεν τηρείται. Εδώ λοιπόν θα σας ζητήσω κατεπηγόντως να λάβετε δράση. Ευχαριστώ πολύ. Το σημείωσα. θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι σε όλα αυτά τα θέματα το Κοινοβούλιο έχει την πρωτοκαθεδρία και θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από το κοινό. Θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή του κοινού σε όλα τα θέματα αυτά. Γιατί θεωρώ ότι ο απλός προλογούμενος δεν θα το καταλάβει αυτό. Και νομίζω ότι αν συμβεί αυτό θα υπάρξει πίεση για να βρούμε πιο γρήγορα μια λύση. Ευχαριστώ. Μπόγκταν Ζόνσα από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι κύριε Επιτρόπε. Είμαι από την Πολωνία και θα μιλήσω πολωνικά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις ε, ερωτήσεις που ετέθησαν πριν. Στη συνάντηση με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, η κυρία Βαντελάιν είπε και παραθέτω «Μεγάλες επενδύσεις θα απαιτηθούν στους τομείς εκείνους που πρέπει να χρησιμοποιήσουν νέα τεχνολογία και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Και γι' αυτό το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει αυτές τις περιοχές. Αυτέ τι περιφέρειε. Τέλο παράθεση. Στην γραπτή απάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο είπατε και παραθέτω ότι βλέπετε την ανάγκη για νομοθετικέ προτάσει όσον αφορά το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την επίτευξη των στόχων για την αλλαγή του κλίματος. Υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη που χρειάζονται καθαρές επενδύσεις. Μπορείτε να πείτε λίγα περισσότερα για αυτό το Ταμείο. Πώς θα κατασκευαστεί, πώς θα οικοδομηθεί και πώς θα γίνει η κατανομή των πόρων. Πώς θα οργανωθεί αυτή η κατανομή των πόρων. Η στοχοθεσία είναι η εξή, επαναλαμβάνω. Οι περιφέρειες που είτε επιβαρύνονται λόγω παραγωγής εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, είτε περιοχές που έχουν βιομηχανίες που εκπέμπουν διοξιδίου του άνθρακα και γι' αυτό είναι υποποίηση, αυτοί να είναι λοιπόν αυτοί που θα έχουν πόρους από αυτό το Ταμείο Δικής Μετάβασης. Και σκοπός ποιος είναι οι βιομηχανίες οι οποίες έχουν υψηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, είτε να αναβαθμιστούν τεχνολογικά προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές, να μηδενιστούν, είτε να αντικατασταθούν από άλλες ε, βιομηχανίες Όπω σα είπαμε, τα απαραίτητα κοινωνικά μέτρα τα οποία προαπαιτούνται, ε, εκπαίδευση κτλ. Και να υπάρξει και άλλο ε, ενεργειακό κλάδο. Θα διαθέσουμε λοιπόν μέτρα προς την κατεύθυνση, μέσα προ την κατεύθυνση αυτή. Και σίγουρα θα υπάρξουν ε, χρηματοδότηση από τα διευθυντικά ταμεία και εγγύησει από τα κράτη-μέλη αν υπάρξουν ε, νομοθεσία από κάποια κράτη-μέλη για να αλλάξουν οι κανόνες ε, επιτόπου σε ό,τι αφορά τις ε, επενδύσεις, νομίζω ότι θα δοθεί κίνητρο για ιδιωτικές επενδύσεις και θα επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή. Θα είναι καταλήτης λοιπόν αυτός σε ό,τι αφορά της εξελίξης στον κλάδο. Επαναλαμβάνω, δεν θα φτάσει από μόνο του το Ταμείο. Δεν θα αρκέσει. Σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης έχουμε ανάγκες σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος. Εκεί θα χρειαστούν παντού λοιπόν επενδύσεις και γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μέσα για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Από το Ταμείο Συνοχής, από τα Δευτερικά Ταμεία, από το Ταμείο Ανάπτυξης Υπέθρου, Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποτυπωθούν στον προγραμματισμό. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τότε καθαρές επενδύσεις. Χαίρομαι για αυτά που άκουσα, για αυτά που μας είπατε. Κάτι άλλο να ρωτήσω. Χθες άκουγα την Ελίζα Φερέιρα που είναι υποψήφια για, στη θέση Επιτρόπου Περιφερειακών Υποθέσεων και αναφέρθηκε σε περιοχές με χαμηλό επίπεδο πληθυσμού, αραιοκατοικημένες, υπέροχα βουνά όπως είναι τα Καρπάθια Φερρυπίν, που είναι στα σύνορα διαφόρων χωρών. Μπορείτε να φανταστείτε υποστήριξη για υποδομές σε περιοχές όπως είναι τα Καρπάθια Όρη ή ο δρόμος που συνδέει βορρά-νότο όπως αυτός που υπάρχει στη Φιλανδία. Τα Καρπάθια έχω υπόψη μου, διότι είναι διασυνοριακή περιοχή όπου χρειάζονται υποδομές. Αυτό θα βοηθούσε να αναπτυχθεί αυτή η υπέροχη γωνιά της Ευρώπης. Αν ναι, θυμάμαι καλά ε, από την εμπειρία μου ε, ως Επιτροπός ε, για την Περιφερειακή Ανάπτυξη αναφέρεσαι στη στρατηγική της Καρπάθια. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Μου δώσατε όμω μία λέξη κλειδί. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα είναι ένα από τα βασικά μας καθήκοντα και κυρίω σε ό,τι αφορά του εκπροσώπου των νέων κρατών μελών, να το πω το εξή. Θα πρέπει να επενδύσουμε στου σιδηροδρόμου και κατά την προετοιμασία του μοραδικού μου χαρτοφυλακίου, αν με βεβαιώσετε, και κατά την προετοιμασία τη ακρόαση, διαπίστωσα ότι, για παράδειγμα, σήμερα η αναβάθμιση του συνδρομοδικού δικτύου για υπερταχείες ε, συνδρομικές οδούς που θα είχαν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν ε, μικρές αποστάσεις ε, αεροπορικές δεν θεωρούνται μέτρο για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Αυτό θα πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί προφανώς και έχει μεγάλη σημασία αν ο κόσμος δεν παίρνει αεροπλάνα και παίρνει τρένα. Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ με πολύ συγκεκριμένα μέτρα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια που πρέπει να επιδείξουμε στον προγραμματισμό και από που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Και νομίζω ότι έτσι θα προκύψουν πάρα πολλά σωστά προγράμματα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο με τους ίδιους κανόνες. Δίνω το λόγο στον κύριο Σιφκρίτ Μουρεσάν για το ΕΛΚ. Α, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Έλενα Κουντουρά, για την ΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω ελληνικά. Κύριε Χαν, η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε για να καλύψει μια συγκεκριμένη ανάγκη να στηρίξουμε τις πιο αδύναμες περιφέρειες, να τις θωρακίσουμε, ώστε να είναι σε θέση να σταθούν ανταγωνιστικά σε μια ενιαία αγορά που δεν γνωρίζει σύνορα. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, λοιπόν, προχωράει εντατικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, η προηγούμενη επιτροπή της οποίας ήσασταν μέλος πρότεινε την περικοπή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχή κατά 10%. Πιστεύετε κύριε Χάνο, ότι η πολιτική συνοχή χάνει το λόγο ύπαρξή τη, και αν όχι πώς θα εξασφαλίσετε ότι τα κονδύλια δεν θα υποστούν περικοπές. Και ένα δεύτερο σημείο, το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι συμβατό με τους κλιματικούς μας στόχους. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι η επίτευξη των κλιματικών μας στόχων θα είναι δίκαιη για όλους και ειδικά για τους οικονομικά ασθενέστερους και για αυτούς που εργάζονται σε τομείς με αυξημένο αποτύπωμα άνθρακα. Πώς θα φροντίσετε μέσω του προϋπολογισμού τις ανάγκες αυτών των ομάδων. Επαρκεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ευχαριστώ. Ως πρώην Επιτροπός Περιφερειακής Ανάπτυξης, είχατε τιμή και τη χαρά να είμαι Λοιπόν, τέτοιο επιτροπό, το... καταρχά δεν είναι 10% η μείωση, είναι μικρότερη, αλλά όλε οι περικοπέ πονών. Αποφασίσαμε στην επιτροπή αυτή, μετά από πολυετής διαπραγματεύσεις, να εξυγχρονίσουμε περαιτέρω το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εδώ λοιπόν Πρέπει να κάνουμε συμβιβασμού, Δεν υπάρχει άλλη λύση. Συμβιβασμού λοιπόν. Αν θέλουμε να ξοδέψουμε παραπάνω χρήματα για την έρευνα, αν θέλουμε να ταπανίσουμε πιο πολλού πόρου για την γειτονία, για να ενισχύσουμε παράλληλα και την Ευρώπη, αν θέλουμε να επενδύσουμε πιο πολύ για την επιτόπιση της αλλαγής του κλίματος, εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνουν ανακατατάξεις. Από την άλλη, έχετε απόλυτο δίκιο που λέτε ότι ο στόχος της πολιτικής ε, συνοχής είναι να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν οι ασθενέστερες ε, περιοχές και περιφέρειες. Εδώ ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν θετικές ε, εξελίξεις και αυτό αποτυπώνεται λοιπόν στον προπολογισμό. Άρα σε τελική ανάλυση θεωρώ ότι ήταν δίκαιη και ισορροπημένη η πρόταση που υποβάλαμε. Και πολλές φορές έχω επισημάνει το δυναμικό του Ταμείου Δίκης Μετάβασης. Και αν θυμάμαι καλά, ε, έχω δύο περιοχές στην Ελλάδα υπόψη, η μία στην Πελοπόννησο, δεν κάνω λάθος, που έχουν αξιοποιήσει και θα αξιοποιούσαν μάλλον το Ταμείο αυτό, αν ε, υπήρχαν συγκεκριμένα προγράμματα και είμαι πεπισμένος και από, από πλευράς της Ελλάδος θα γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις, έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα δαπανηθούν τα μέτρα αυτά για να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Συμπληρωματική. ήθελα τώρα να σταθώ στο σημαντικό ζήτημα του τουρισμού. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός ο τουρισμός που είναι πυλώνας της οικονομίας και καταλήτης για την ανάπτυξη πολλών παραγωγικών κλάδων και αποτελεί το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, στηρίζει εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ειδικά σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές που δεν έχουν διέξοδο σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επιτακτικά την ένταξη του τουρισμού στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο με ένα ποσό μάλλον συμβολικό που απέχει πολύ από τις πραγματικές ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές για να αποφεύγουμε παρανοήσεις δεν είναι η χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες άλλωστε έχουν πρόσβαση σε άλλα ευρωπαϊκά ταμεία. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού και ένα μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων προορισμού σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, ζητημάτων ασφαλείας που έχουμε ζήσει πολλές τα τελευταία χρόνια και άλλες ανθρωπογενείς κρίσεις όπως το προσφυγικό αλλά και για τη διάσωση χιλιάδων θέσεων εργασία σε περιπτώσεις καταστροφής τουριστικών κολοσσών. Αναγνωρίζετε κύριε Χάν τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία και την απασχόληση. Δεσμεύεστε ότι θα στηρίξετε την ένταξη του τουρισμού στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Also, um, Όπως και εσείς είμαι και εγώ από μια χώρα που έχει να κάνει πολύ με τον τουρισμό. Και ζει σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Έχετε και για δεύτερη φορά απόλυτο δίκιο. Ε, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος τομέας εσόδων ο τουρισμός στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να συνεχίσουν τα πράγματα να πάνε καλά στον τουρισμό. Στον τουρισμό λοιπόν έχουμε διάφορες πολλαπλές προκλήσεις. Έχουμε προορισμούς ε, που παραπονιούνται ότι έχουν υπερβολικά πολλούς τουριστές. Το θέμα είναι να υπάρχει και μια βιώσιμη λοιπόν προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον τουρισμό μας. Έχουμε και τα συμφέροντα των πολιτών μας εδώ, τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα, ήμουν και ιδιαίτερα α, ταγμένο στο θέμα αυτό ως Επιτροπός. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό. Αλλά ο τουρισμός δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα από πλευρά τη πολιτική ε, υποστήριξη όμω και χρηματοδότηση είναι κάτι όπου τα μέσα, τα δραστηριοτικά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Και θυμάμαι για παράδειγμα στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν σημαντικά ποσά για τουριστικούς προορισμούς προκειμένου να δημορφωθούν με βιώσιμο τρόπο και να καταστούν ελκυστικοί. Αυτό έγινε και θα συνεχίσει να γίνεται στο μέλλον αν τα μεμονωμένα κράτη-μέλη το επιθυμούν. Εμείς θα επιμείνουμε στο εξή. Οι επενδύσεις στον κλάδο αυτό να συνδέονται και πάλι με τους στόχους για το κλίμα. Εδώ υπάρχουν αναρρύθμιτες δυνατότητες να διαμορφώσουμε τις επενδύσεις αυτές με έξυπνο τρόπο. Thank you. Ευχαριστούμε. Πράγματι όμως τώρα περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μούρεσαν όμως, Παρακαλώ, σημειώστε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας, γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Να τηρείτε ένα λεπτό ερώτηση, ένα λεπτό απάντηση. Ο κύριος Μουρισάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εφόσον επιβεβαιωθείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσείς θα αναλάβετε ηγετικό ρόλο όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα επόμενα 7 χρόνια. Έχουμε ακούσει πολλά για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, τώρα για τον ετήσιο προπολογισμό. Η εμπειρία μα δείχνει ότι το Συμβούλιο ποτέ δεν είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί με το Κοινοβούλιο παρά μόνο τι τελευταίε ημέρε τη ε, διαδικασία. Κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην όλη διαδικασία και δημιουργεί και την εντύπωση στον έξω κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε το 2018 που ήμουν εγώ γενικό εισηγητέ για τον προπολογισμό, αλλά αντιστάθηκε το Συμβούλιο. Ρωτώ λοιπόν, εσείς θα μπείτε στον αγώνα με το Συμβούλιο προκειμένου να έρχονται πιο νωρί στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και από την εμπειρία που έχετε ως υπουργό, τι χρειάζεται για να πετύχει αυτό. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι ότι όταν διαφέρουν οι απόψεις ε, της Επιτροπή, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίξει το ρόλο του δεύτερου διαπραγματευτή. Κατά το παρελθόν, ε, τα τελευταία χρόνια, ακούσαμε διαφορετικά πράγματα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προκειμένου να ε, ευχαριστούμε το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο ανάλογα. Εσείς τι θα κάνετε, θα το αποφύγετε αυτό, να λέτε άλλα στον ένα και άλλο στον άλλον. Θα κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά και θα προσπαθήσω να είμαι ουδέτερος διαμεσολαβητής, να διευκολύνω λύσεις, να καταφέρνω λύσεις. Συνήθως υπόσχομαι λιγότερα και καταφέρνω περισσότερα. Κατά κάποιο τρόπο αυτή θα είναι η προσέγγιση μου και τα επόμενα ε, πέντε χρόνια. Και συμφωνώ απόλυτα και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη δυσαρέσκειά σας. Δεν την έχω ζήσει από πρώτο χέρι, αλλά κοιτώντα τα διάφορα έγγραφα και τις διάφορες εκθέσεις, πραγματικά δεν είναι ικανοποιητική αυτή η κατάσταση. Να έχουμε ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο δεν χρησιμοποιείται μέχρι την τελευταία στιγμή και μόνο την τελευταία στιγμή ξαφνικά ε, μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κοιτάξω να το αποφύγω. Να έχουμε εκ των προτέρων διάφορες συναντήσεις και να πιέζω για συναντήσεις και όχι μόνο να προσπαθήσω επίσης να εντοπίσω τα τεχνικά ζητήματα τα οποία μπορούν εύκολα και γρήγορα να επιληθούν και να αφήσω τα πιο, πώς να το πω, πολιτικά ζητήματα, τα οποία επίσης μπορούν να λυθούν βέβαια πιο γρήγορα, ώστε να καταλήξουμε μόνο σε δύο-τρία κέρια ζητήματα, τα οποία φαίνεται ότι αποτελούν μια δυσκολία είτε για το Συμβούλιο είτε για το Κοινοβούλιο προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν οι τρεις εβδομάδε και οι τρεις για την επίτευξη συμφωνίας. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα τα καταφέρω, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Γιατί μια τέτοια κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική ούτε για μένα, ούτε για τους συνεργάτες μου, αν έχουμε την ίδια κατάσταση που πρέκυψε πέρυσι, για παράδειγμα. Συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο πάλι θα υπάρξουν πληρωμέ προς τους δικαιούχου που θα μας έχουν μείνει από το προηγούμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία προχωράμε και ότι έχουμε με την συνοχή. Οπότε τελικά θα υπάρξουν πολύ καθυστερημένοι λογαριασμοί που δεν θα μπορούμε να τους πληρώσουμε. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις αρνητικές επιπτώσεις ενό ε, τέτοιου όγκου καθυστερημένων πληρωμών και επίσης από τη δικιά σας εμπειρία από την περιφερειακή πολιτική κύριε Επιτροπέ, τι μαθήματα έχουμε πάρει ώστε στην αρχή της ε, του του δημοσιονομικού πλαισίου να γίνεται πιο γρήγορα η απορρόφηση, ώστε να μην μας μείνουν όλοι οι λογαριασμοί προς πληρωμή στο τέλος της περίοδου. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο. Χάρη στο Κοινοβούλιο και τις σκληρές διαπραγματεύσεις που κάνατε την τελευταία φορά, εισάγατε την ευελιξία. Και αυτή η ευελιξία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, σε περίπτωση τέτοιων δυσκολιών ε, στις πληρωμές. Δεύτερον, αυτό που είπατε είναι άλλη μια απόδειξη, άλλο ένα παράδειγμα που δείχνει ότι χρειαζόμαστε γρήγορα συμφωνία επί του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Την προηγούμενη φορά το γεγονός ότι η απόφαση λήφθη μόνο δύο εβδομάδες πριν την εκπνοή οδήγησε στο λεγόμενο backlog, δηλαδή στους καθυστερημένους λογαριασμούς που έπρεπε να πληρώσουμε και είχαμε τα διάφορα ατομικά προγράμματα αλλά και τις καθυστερήσεις. Συνεπώς και γι' αυτό πιέζουμε κι εμείς όσο πιο γρήγορα μπορούμε να μπούμε στην υλοποίηση τόσο το καλύτερο, γιατί έτσι θα καταφέρουμε καλύτερα τους πολιτικούς μας στόχους. Είναι άλλο ένα παράδειγμα που δείχνει ότι πρέπει να πιέζουμε και να είμαστε επικεντρωμένοι όσο γίνεται περισσότερο στην υιοθέτηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Κύριε Γκουαλμίνη τώρα, Σοσιαλδημοκράτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Χάν. Πάω στο θέμα τη αναθεωρήσεω των ιδίων πόρων. Ήδη μιλήσατε γι' αυτό. Όπω καταλαβαίνετε όμω αυτό είναι σημαντικό θέμα για μα, Η Ursula von der Leyen, εκλεγή σαν πρόεδρο τη κατευθείαν γραμμέ, αναφέρθηκε στο ψηφιακό φόρο που θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στους στόχους της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δίκαιης φορολόγησης και το νέο φόρο για τον, το άχθος του άνθρακα και επίσης ο ψηφιακός φόρος μπορεί να συνδεθεί με το CCCBT για τις πολυεθνικές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας. Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι ίδιοι πόροι θα μπορούσαν να προσθεθούν στο φάσμα των ιδίων πόρων που ήδη έχουν σκιαγραφηθεί και προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και ένα χρόνο. Απάντηση. Θα μπορούσαν και θα έπρεπε να προσθεθούν. Αυτό που έχω διαισθανθεί μέχρι τώρα και αυτά που άκουσα και αυτά που διάβασα μου δείχνουν ότι υπάρχει ανοιχτή στάση όσον αφορά το διασυνοριακό φορά άνθρακα. είναι μια ιδέα που ακούγεται στην Ευρώπη από διάφορες πηγές. Πολλοί είμαστε θετικοί όσον αφορά αυτό. Πρέπει να διερευνήσουμε πώς μπορεί να δομηθεί, να διαρθρωθεί αυτή η προσέγγιση και πώς να υλοποιηθεί. Άρα, διάκειμε θετικός. Όπως είπα και σε προηγούμενη απάντηση για τον ψηφιακό φόρο, Υπάρχουν πολλοί δισταγμοί σε κάποια κράτη-μέλη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να παραιτηθούμε. Θα ήταν άδικο αν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και κοιτάζω προς τον κύριο το φίλο μου θα ήταν άδικο εάν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να ξεφύγουν. Ίσως θα έπρεπε να επανακαθορίσουμε μια ενδεχόμενη προσέγγιση, το ώστε να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες. Όμως δεν πρέπει να παρετηθούμε. Αν μπορούμε να μαζέψουμε χρήματα από αυτή την πηγή, βεβαίως αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σε διάφορες πρωτοβουλίες για το κλίμα, να διατεθούν αυτοί οι πόροι. Διευκρινιστική ερώτηση. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Για τους ιδίους πόρους και πάλι είναι περισσότερο θέμα κουλτούρας αν θέλετε. Αν μπορέσουμε να θεσπίσουμε ευρωπαϊκά, πραγματικά ευρωπαϊκούς ιδίους πόρους με συνεισφορά από τα ΕΠ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλλαγή νοτροπίας, εξευρωπαϊσμό της δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν πρέπει να πούμε στα κράτη-μέλη, κοιτάξτε, θέλουν περισσότερα χρήματα από εσά γιατί αν το πούμε αυτό δεν θα επανεκλεγούμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα νοτροπία, να έχουμε έσοδα που σχετίζονται στενά με τις πολιτικές προτεραιότητες των νέων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα έχουμε θητεί αυτά τα πέντε χρόνια. Ερώτηση. Θα συνεργαστείτε στενά με το Συμβούλιο για να προωθήσετε με τέτοια προσέγγιση και εκτιμώ το συσχετισμό που κάνετε στην παρουσίασή σας μεταξύ της αναθεωρής των ιδίων πόρων και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τις σχετικές διαπραγματεύσεις για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Απάντηση. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Σε έναν ιδεώδη κόσμο θα πρέπει σταδιακά να αυξάνουμε το ποσοστό των ιδίων πόρων στο γενικό προπολογισμό. Δεν πρέπει να ειδωθεί αυτό σαν ένα είδος αστιστάθμισης θα πρέπει να είναι αύξηση συμπληρωματική και να μειωθεί η εισφορά από το ΑΕΠ από τα κράτη-μέλη στο Γενικό Προπολογισμό. Αλλά υπάρχει και άλλος λόγος για τον οποίο είμαι τόσο πολύ υπέρ των ιδίων πόρων. Όχι από πλευράς οικονομικής και μόνο. Πώς να το πω τώρα. Και από πλευράς νοοτροπίας ή στην ατμόσφαιρα που επικρατεί. Θέλω να ξεπεράσουμε αυτό το διχαρισμό μεταξύ εκείνων που συνεισφέρουν ξεκαθάρα και εκείνων που είναι καθαρά δικαιούχοι. Στη χώρα μου 95% φόρων και εισφορών συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο και διάφορες περιοχές δεν, δεν ξέρουμε δηλαδή πραγματικά αν παίρνουν ή δίνουν χρήματα οι περιφέρειες. Θα ήταν ιδεώδες αν καταλήξουμε και στην Ευρώπη σε ένα τέτοιο επίπεδο, δηλαδή όπου δεν κάνουμε διαφοροποίηση. Ο κ. Έτιγκερ, ο παρόν επίτροπο για τα θέματα του προπολογισμού, λέει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ δικαιούχων και εκείνων που συνεισφέρουν δεν ισχύει όπως περιγράφεται ακριβώς. Πολύ συχνά ωφελούνται αυτοί που δίνουν χρήματα από επενδύσεις σε χώρες δικαιούχους. Υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Ευχαριστούμε. Ολιβιέ Σαστέλ, τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ από το Ρινιού. Στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στο σεβασμό του κράτους δικαίου. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εξάλλου μέσα για την καλή εφαρμογή των αξιών της. Όμως δεν υπάρχει καμία άμεση αντίδραση και αποτελεσματική σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξάλλου πρότεινε στα πλαίσια του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου έναν ειδικό μηχανισμό προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένης αδυναμίας όσον αφορά το κράτος δικαίου σε κάποια χώρα, χωρίς να μιλάει για οικονομικές κυρώσεις. Εσείς μιλάτε για την προστασία του προπολογισμού της Ένωσης. Εσείς δεσμεύεστε να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμό αυτό, ο οποίος ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε τέτοιες παραβιάσεις μιας χώρας και δεδομένου ότι πρέπει με συναπόφαση να εγκριθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, εσείς τι θα κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κατά τη γνώμη σας για την υιοθέτηση αυτού του μέτρου. Τέλος, δεδομένου ότι ο μηχανισμός αυτός διαρθρώνεται γύρω από ε, βασικά άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού, εσείς Πώς προβλέπετε αυτή τη διάρθρωση, δηλαδή για το άρθρο 61, σύγκρουση συμφερόντων και το 63, 8 και 91 όσον αφορά την ε, πάυση πληρωμών σε περίπτωση σοβαρών αδυναμιών. Σε ό,τι αφορά το χρηματοοικονομικό κανονισμό, Έχουμε το άρθρο 61. για το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο το 2018. Δημιουργείται λοιπόν η δυνατότητα όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων να υπάρχει δυνατότητα διορθώσεων, χρηματοοικονομικών διορθώσεων. Αλλά σε πρώτη σε πρώτο επίπεδο έχουμε την ιδέα εισαγωγή ενός μηχανισμού για το κράτος δικαίου. Αν όμως έχουμε α, τα ασταλείε στο θέμα του κράτους δικαίου σε κάποιο κράτος μέλος, δεν, δεν την τακτική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Τότε λοιπόν μπορεί να οδηγηθούμε σε διαδικασία επί παραβάση. Αυτό δεν είναι τιμωρία, είναι προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Αν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Να γίνονται λοιπόν, να υπάρχει δυνατότητα χρηματοοικονομικών διορθώσεων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν υπάρχουν προβλήματα, ελλείψεις, σε ό,τι αφορά την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας. Αν τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο μηχανισμός, θα μπορούμε στο μέλλον να αναλάβουμε δράση, γιατί ένα τμήμα των ε, φόρων προστιθέμενης αξίας θεωρώ ότι είναι στο προϋπολογισμό ως ήδη πόροι. Αν υπάρχουν δυσκολίες ή προβλήματα σε ό,τι αφορά την επιβολή επιχειρηματικού φόρου, δεν θα έχουμε δυνατότητα ε, επέμβασης γιατί, παρέμβασης, γιατί αυτό δεν αφορά ευρωπαϊκούς πόρους. Αν λοιπόν υπάρχει ευρωπαϊκή ε, εμπλοκή, ευρωπαϊκή πόρη, εκεί θα έχουμε ε, δυνατότητα παρέμβασης. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ για την ε, απάντησή σας. Δεν άκουσα τίποτα όμως για το χρονοδιάγραμμα ε, λειτουργίας αυτού του νέου μέτρου, του νέου κανονισμού. Αλλά έχω και συμπληρωματική ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα ε, θέσει σε εφαρμογή αυτόν τον νέο κανονισμό, ενώ συγχρόνω θα πρέπει να ετοιμάσει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των διαφόρων διευθύνσεων, ρέγγιο, απασχόληση κτλ. και να αναλάβει από μόνη τη τον ρόλο εντοπισμού των αδυναμιών των χωρών μελών. Εσείς θα συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Όλαφ, την Europol, Eurojust κτλ. Για να υπάρχει κάποια συνοχή και να συνδέσουμε όλα αυτά τα θέματα με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, υποθέτω ότι αναφέρεστε ότι αναφέρεστε στο γεγονός ότι στον κανονισμό αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα ρυθμιστούν όλα αυτά στα πλαίσια ενός κανονισμού και να μην γίνουν τμήματα των διαπραγματεύσεων πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το καταφέρω αυτό. Γιατί όντως πρόκειται για κάτι ξεχωριστό. Αυτή υπαρκτό. Που δεν ισχύει μόνο για το επόμενο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, ξεπερνά το επόμενο πλαίσιο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ο κοινό μα σκοπό και αυτό θα πολεμήσουμε να πετύχουμε. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο στοιχείο. Συνεργαζόμαστε στενά με τον Όλαφ. Ο Όλαφ λοιπόν και ε, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάνω από 500 στον αριθμό. Σχεδόν 400 και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί λοιπόν έχουν ε, καθήκον να κοιτάξουν τα θέματα αυτά. Μόλι μου τελείωσε και ο χρόνο ομιλία μου όμως και θα απαντήσω κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Βίντσιχ, η Αγγέλικα Βίντσιχ από το ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Μα αναφέρατε το δύσκολο χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά το πουδουπού κάθε περαιτέρω καθυστέρηση ουσιαστικά υπονομεύεται συμφωνία για να μην επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εμείς από το Κοινοβούλιο, ακόμα και από χρονική πίεση, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε ένα κακό σεμιβασμό. Αν δεν υπάρξει λοιπόν συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τι γίνεται υπάρχει δυνατότητα παράτασης. Ε, εφόσον όμως υπάρχουν σε λειτουργικό επίπεδο και σε νομοθετικό επίπεδο οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο ζητά ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι πιστεύετε για αυτό το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αν είστε υπέρ αυτού θα δεσμευτείτε να περάσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουμε εγκαίρως να καταρτήσουμε ένα τέτοιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι στη συζήτηση προέκυψε αυτό. Ότι θα πρέπει να έχουμε όλοι στην καρδιά μας ε, την πιο γρήγορη δυνατή επίτευξη συμφωνίας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να ακολουθήσουμε τους πολιτικούς μας στόχους, τον εξυγχρονισμό του προπολογισμού κτλ. κτλ. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν επίσης και καθυστερήσεις στην εφαρμογή. Εκεί θα εστιαστούμε. Να πω επίση ξεκάθαρα το εξή. Προφανώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και οι αντίστοιχε ε, υπηρεσίε θα πρέπει να έχουν ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τη συμφωνία αυτή εγκαίρω. Μία πρόταση από πλευράς μας όμως θεωρώ ότι θα κινητοποιήσει όλη την ε, διαθεσμική μηχανή. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο θα κληθούν ε, να τα εξετάσουν αυτά γιατί αποτελεί αυτό που πρόταση νομοθετική. Και αυτό θεωρώ ότι θα αποτρέψει την προσοχή μας από τον πραγματικό στόχο, την επίτευξη της συμφωνίας. Στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη-μέλη. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτό. Αλλά σας υπόσχομαι ότι αν χρειαστεί, εάν παραστεί ανάγκη, θα υποβάλουμε σχετική πρόταση. Αλλά τονίζω ότι αν το συζητήσουμε αυτό τώρα, στην παρούσα χρονική φάση, θα αφαιρέσουμε πίεση για την επιτεύξη των διαπραγματεύσεων. Και αυτό θεωρώ ότι δεν συμφέρει κανέναν τονίζω το εξή, ότι κάθε καθυστέρηση στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο σημαίνει καθυστέρηση και στην υλοποίηση των κοινών, φαντάζομαι, πολιτικών μα στόχων. Διευκρινιστική ερώτηση. Το Κοινοβούλιο ζητάει στο μέσα της πολιτικής δημοσιονομικού πλαισίου να γίνει η αναθεώρηση, η υποχρεωτική αναθεώρηση σε ό,τι αφορά το midterm αυτό, revision προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη ε, ανάγκες οι οποίες θα, θα παρουσιαστούν στην πορεία. Θα υποστηρίξετε λοιπόν αυτή τη διάμεση αναθεώρωση και τι θα προτείνετε συγκεκριμένα αν ε, κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα δεν ε, δείξουν ότι έχουν επιτυχία ή δεν πετυχαίνουν το στόχο που έχουν ξεκινήσει για την ενδιάμεσα αναθεώρηση θα είμαι πολύ σύντομο. Απόλυτη υποστήριξη πάντα υπήρχε και θα ξεκολουθήσει να υπάρχει γιατί έχει νόημα. Και αυτό που επίσης έχει νόημα από δική μου πλευρά είναι όλοι μας να δώσουμε την απαραίτητη ευελιξία και να μην περιμένουμε απαραίτητα την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αν δούμε πιο νωρί ότι κάποια προγράμματα δεν απορροφούν τα κονδύλια όπω πρέπει, δεν πετυχαίνουν του στόχου που χρειάζεται, θα πρέπει να κοιτάξουμε και του δείκτε μα, γιατί σε κάποιε περιπτώσει ούκαν το πολλό το F. Και να υπάρξει λοιπόν και πριν την ενδιάμεση αναθεώρηση ενδεχομένω προσαρμογή και ευχαριστώ ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο ήδη για την υποστήριξη τη πρόταση μεγαλύτερη ευελιξία και σε ό,τι αφορά το πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο. Μίσλαβ Κολακούσιτ, μία εγγεγραμμένο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χάν, λέει ο κύριο Κολακούσιτ. Την τελευταία δεκαετία ήσασταν επίτροπος με δύο διαφορετικά χαρτοφυλάκια ένα από αυτά ήταν η περιφερειακή πολιτική. Το άλλο ήταν η διεύρυνση. Τώρα έχετε προταθεί να αναλάβετε ως επίτροπος σε τρίτη θητεία υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι είσαστε ο σωστός άνθρωπος μπορεί να μας δώσει απάντηση στην κάτωθη ερώτηση. Τι θα κάνετε ούτως ώστε να εξασφαλίσετε το ότι οι πόροι από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα διανέμονται ε, πιο ε, δίκαια στα κράτη-μέλη. Να δώσω κάποια παραδείγματα. Το 2014 μέχρι το 2018, δηλαδή τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ρουμανία και η Ουγγαρία είχαν πλεόνασμα 22 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Πολωνία πλεόνασμα 51 δις ευρώ. Η δημοκρατία της Κροατίας, αν συγκρίνουμε με αυτές τις χώρες, έχει λάβει 12 φορές λιγότερα χρήματα. Με άλλα λόγια, 28 φορές λιγότερα χρήματα από την Πολωνία. Εδώ βλέπουμε κάποια ποσοστά, κάποιες αναλογίες από 0,5 μέχρι δεκαπλάσιους πόρους που έχουν λάβει κάποιες χώρες δικαιούχες εν συγκρίση με τις εισφορές τους. Και δεν νομίζω ότι αυτό ε, οφείλεται στο ρυθμό απορρόφησης. Η Ιρλανδία, Φερρυπίν, είχε πολύ περισσότερα χρήματα που έλαβε και αργότερα ήταν σε αρνητικό πρόσημο το ισολογισμός της. Ε, Η συζήτηση αυτή μου είναι ιδιαίτερα γνώριμη. Και έχω και κάποια αριθμητικά στοιχεία κατά νου, γιατί Είχα πριν από μία εβδομάδα τον Πρωθυπουργό σα ε, σε επίσκεψη και ο οποίο μου παρουσίασε το θέμα αυτό. Η διανομή των ταμείων, ε, των ευρωτικών ταμείων, αυτό αναφέρεται ουσιαστικά. Αυτό γίνεται με μία μέθοδο υπολογισμού περίπλοκη, λιγότερο περίπλοκη, κατά Πρώτον, 85% βασιζόμαστε στο, σημείο, στο επίπεδο διαβίωσης ε, των ε, υπαλλήλων, των απασχολούμενων. Αυτή είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ύστερα, σε μικρότερο ποσοστό έχει να κάνει και η απορρόφηση μεταναστών ή όχι. Και όλα αυτά λοιπόν καταλήγουν σε ένα συντελεστή που έχουν που σχετίζεται με το επίπεδο διαβίωσης, βασιζόμενη και σε στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Εν πάση για να μην λόγο... όλοι καλούνται να κάνουν περικοπές, φανταζόμαστε. Γιατί, γιατί οι χώρες αυτές, όταν φτάσουν στο επίπεδο στόχο, που ήταν να υπάρξει μια εξισορρόπηση με το επίπεδο διαβίωσης. Η Κροατία, να σας πω για παράδειγμα, εξακολουθεί, μάλλον πλέον συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ταμεία πως ποσοστό μάλλον ανάθεσης ε, ε, διαφορετικών ταμείων ε, στη δεύτερη τρίτη θέση νομίζω είναι σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την, ε, τα έσοδα που λαμβάνει κατά κεφαλή, κατά κεφαλή σε ό,τι αφορά τα διευθυντικά ταμεία. Όλα αυτά λοιπόν να τα έχουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για ίση κατανομή. Σας ευχαριστώ. Έχω μια σύντομη ερώτηση. Είναι μια Ερώτηση επί της αρχής. Συμφωνώ προσωπικά ότι περιορισμός σε δύο θητείες για πολιτικά καθήκοντα που δεν αποτέλεσματα εκλογών αυτές, αυτοί οι διορισμοί θα πρέπει να είναι κάτι που αρκεί οι δύο θητείες. Δύο θητείες πρέπει να αρκούν και τώρα είστε υποψήφιος για τρίτη θητεία. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε περιορισμό αριθμού θητιών, να περιορίζεται σε δύο θητείες υπηρεσία ή μπορείτε επαόριστον να είστε επίτροπος, να είναι κάποιος επίτροπος. Äh, δεν σκοπεύω να αναμειχθώ σε αυτή τη συζήτηση. Ε, είμαι εδώ υποψήφιος για τρίτη φορά. Δέχθηκα να, προς τη χώρα μου να επιτελέσω το ρόλο αυτό και νομίζω ότι στην πολιτική δεν είναι ε, κακό να έχει κανείς ε, σημαντική εμπειρία και όπως βλέπετε πέντε χρόνια ε, σημαίνουν μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερη γνώση η οποία σε τελική ανάλυση ωφελεί τον κόσμο. Και όπως και εσείς ξέρετε και πολλοί κόσμος ξέρει μπορεί να δει ο καθένας πώς τα πήγε ο υποψήφιος όταν υπάρχει διαφάνεια σε την αφορά την απόδοση. Γιατί κάποιο ο οποίο έχει η πολιτική εμπειρία, έχουμε μια καλύτερη εικόνα, εν πάση περιπτώσει, από κάποιον που δεν έχει ασκήσει τα καθήκοντα αυτά. Αν λοιπόν ο, ο υποψήφιος έχει δέσμευση και θέλει να υπηρετήσει, να, να ασκήσει το ρόλο του αυτό, δεν βλέπω ότι πρόβλημα υπάρχει. Η κυρία, κυρία Μόνικα Βάνα, εκ μέρου των Πρασίνων. Κύριε Πίτροπε, γνωριζόμαστε από την Βιέννη. Οπότε δεν σας εκπλήξει η επόμενη ερώτησή μου για την ισότητα των δύο φύλων και τη συνεκτίμηση της διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Λοιπόν, στην κοινή δήλωση όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, βλέπουμε ότι δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος. Δεν έχουμε στρατηγική για την ισότητα ε, και δεν υπάρχουν καν στοιχεία, δεδομένα, ε, κατά φύλλο και δεν έχουμε καν και αξιολόγηση αντικτύπου για τον προπολογισμό ανάλογα με το φύλλο. Στις γραπτές τώρα ε, απαντήσεις σας είπατε πόσο πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ισότητας, αλλά δεν μας λέτε με ποιον τρόπο πιο συγκεκριμένα θα υλοποιήσετε τις προθέσεις σας την επόμενη πενταετία. Οπότε ρωτάω συγκεκριμένα τι βήματα θα αναλάβετε ώστε να υπάρχει η χρηματοδότηση αυτή εξίσου και για τα δύο φύλλα και να υπάρχει για τον προπολογισμό αυτό ο κατάλληλος έλεγχος και εποπτεία. Απάντηση. Πρέπει να ομολογήσω. Αν μιλάτε, για παράδειγμα, για τον μελλοντικό τίτλο 7, Δίκηση, είναι πιο εύκολο για μας όλα αυτά να τα κοιτάξουμε και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι γιατί είναι κάτι που έχει να κάνει με μας. Όπως είπα, 80% του προπολογισμού μας δαπανάται με κοινή διαχείριση, επιμερισμένη διαχείριση με τις χώρες μέλη. Αντιλαμβάνομαι τον σκεπτικισμό σας. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το ζήτημα. Και είναι σημαντικό ε, στην αξιολόγηση αντικτύπου που κάνουμε να λάβουμε υπόψη μας και στοιχεία που έχουν να κάνουν ε, με τα δύο φύλλα για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στις πολιτικές μας. Επίσης, στο πλαίσιο για τις επιδόσεις μας, πρέπει και εκεί να δούμε συγκεκριμένους δείκτες που να μας δείχνουν πού βρισκόμαστε. Τώρα όμως, πρέπει να δούμε αναπολιτική τι θα κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε όλα να τα δούμε με τον ίδιο τρόπο και να κάνουμε τα ίδια για τα πάντα, αλλά θέλω πάρα πολύ να έχουμε συνολικά δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εντύπωση του πού βρισκόμαστε και ανάλογα να εφαρμόσουμε ό,τι χρειάζεται για την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα μέσω του προπολογισμού, μέσω των εταίρων μας, μέσω των πολιτικών μας κτλ. Πάνω σε αυτό πρέπει να εργαστούμε περισσότερο πράγματι. Και καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έρθω να συνεργαστώ μαζί σας δεν ξέρω με άτυπους τρόπους ε, επίσημους προκειμένου να προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε τι μέτρα θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Εγώ πάντως συμφωνώ ότι έχουμε καθυστερήσει, ότι είμαστε πίσω, αλλά έχει να κάνει με την πολυπλοκότητα του τρόπου με τον οποίο δαπανώμε τα χρήματα. Και το ότι πρόκειται για επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη-μέλη. Συμπληρωματική, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την απάντησή σας και που λέτε ότι θα τα ξαναπούμε για να προχωρήσουμε. Και ευχαριστώ που αναφέρατε και το προσωπικό, γιατί πράγματι το χαρτοφυλόκιά σας είναι προπολογισμό και δίκηση. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κεφάλαιο για την ποικιλομορφία και προκειμένου να υπάρχει χώρο εργασία καλός για όλου, για όλε τι κατηγορίε ανθρώπων, άντρε γυναίκε, ΛΟΑΤΚΙ κλπ, κλπ. για ολόκληρο το προσωπικό, κάθε κατηγορία. Εσεί, λοιπόν τι δραστηριότητε προβλέπετε για την επόμενη πεντετία προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτελέσει ένα χώρο εργασία στον οποίο όλοι έχουν θέση μέσα και οι ΛΟΑΤΚΙ και ανεξάρτητα από την σεξουαλική προτίμηση του καθενό. Απάντηση. Αν έχετε 30.000 ανθρώπους υπαλλήλου, ε, προφανώς και υπάρχουν πάντα περιπτώσεις και θα υπάρχουν πάντα περιπτώσεις ακόμα και αν δεν μας αρέσει. Αν δω την ε, ετήσια έρευνα ικανοποίηση του προσωπικού μας, η ικανοποίηση αυτή είναι μεγάλη. Βέβαια, η κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αν κάτι δεν πάει καλά σε μία περίπτωση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Έτσι κι όμως είναι ένα θέμα στο οποίο προχωράμε. Πρέπει να επιδεικνύουμε ευαισθησία. Έχουμε στρατηγική, έχουμε σημεία επαφής για τους ΛΟΑΤΚΙ και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα άτομα με αναπηρίες προκειμένου να μπορούμε να τα βοηθήσουμε. όταν φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αν ας πούμε κάποιος από το προσωπικό έχει παιδιά με αναπηρίες και εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε επιπλέον το προσωπικό. Πάντως η έκθεση έρευνας ε, για το επίπεδο ικανοποίηση του προσωπικού, εκεί βλέπουμε ότι η ικανοποίηση είναι μεγάλη. Πάντα όμως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ακόμα. Ευχαριστούμε Κλωτίτ Αμά Ρινιού. Παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, επανέρχομαι επί του Ταμείου Μετάβασης για να καταπολεμήσει χώρες οι ανατολικές ε, την αλλαγή του κλίματος. Υποστηρίζεται αυτό το θέμα, πολύ καλό. Ε, και παρόλα αυτά έχουμε, έχουμε διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην Ευρώπη. Αν δείτε το, τι γίνεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων και των, και εκπομπών. Η Δυτική Ευρώπη είναι στο κόκκινο, ενώ η Ανατολική στο πράσινο. Λοιπόν, Πώ θα γίνεται η χρηματοδότηση αυτού του ταμείου δικιάσματα, βάση μιλήσατε για προσαρμογή, για διεθνωτικά ταμεία. Δεν ξέρω αν ξέρετε πολύ καλά πώ χρησιμοποιούνται αυτά τα διεθνωτικά ταμεία για ε, θεσμό των υδάτων για υποδομέ βασικές. Θα ήμασταν πολύ ευτυχεί αν υπήρχε μεταξύ Ευρώπη της Δύσεως και του Βουκουρεστίου μία ένας αυτοκινητόδρομος, αν υπήρχε σιδηρόδρομος που να πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάτε με τοπικό τρόπο. Δεν έχετε επαφή με την πραγματικότητα αν μιλάτε για σιδηροδρόμους υψηλή ταχύτητα. στα ιδιωτικά ταμεία για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία μαζί για 7 χρόνια δεν θα αρκούσαν για να χρηματοδοτηθεί ένα σιδηρόδρομο υψηλή ταχύτητα από το Βουκουρέστι στα σύνορα και δεν θα ήταν αποδοτικό από ιδιωτικό τομέα χρηματοδότηση. Κύριε Χάν, θα βρείτε χρήματα, νοπά χρήματα για τις κλιματικές προκλήσεις στην Ανατολή ή ε, θα, τελικά θα παίρνετε τα, τα, τα ρούχα του μιανού για να τα δίνετε στον άλλον, θα μεταφέρετε πόρους από το ένα ταμείο για να τα δίνετε αλλού. Να σας πω πώς ήρθε το 2010 εδώ. Είδα ένα προπολογισμό για ανανεώσιμες ενέργειες και διαπίστωσα ότι ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, το λέω ειλικρινά και στη βυτική Ευρώπη, δεν είχαν εκτελεφθεί τα ποσά αυτά. Έκανα λοιπόν ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο επισκέψεις προκειμένου να υπάρξει απορρόφηση των κονδυλίων αυτών. Να σας πω ότι πέντε χρόνια αργότερα και στα νέα κράτη-μέλη άλλαξε λίγο η νοοτροπία και η προθυμία, για παράδειγμα, να επενδύσουν στην ενεργειακή αποφατικότητα σε ό,τι αφορά τη θερμική μόνωση, για παράδειγμα, θερμομόνωση των σπιτιών, ε, αυξήθηκε δραματικά. Γιατί ε, έγινε κατανοητό ότι το θέμα δεν ήταν μόνο η προστασία του κλίματο, ότι όποιο τελικά ζει ε, σε σπίτια με κακή μόνωση, που είναι συνήθω άνθρωποι λιγότερο τυχεροί, όταν μειώνουν τελικά το λογαριασμό του. τελικά αυτό αποτελεί και κοινωνική κοινωνικό μέτρο. Είναι ένα τομέα όπου δημιουργούνται και θέσει απασχόληση. Είσαστε από τη Γαλλία. Εδώ έχουμε πολύ καλέ εμπειρίε σε ό,τι αφορά τη θερμομόνωση πριν από κάποια χρόνια, το κύμα θερμομόνωση που δημιουργήσε θέσει απασχόληση. Υπάρχουν λοιπόν καλά παραδείγματα. Και σε εμά, ε, από εμά επαφείεται να αποφασίσουμε πόσο θα προγραμματίσουμε τα μέσα αυτά και πόσο αυστηροί θα είμαστε, άκαμπτοι σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητές μας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στον τομέα του κλίματος, υπάρχει και η διάσταση εξή. Η επεξεργασία λιμάτων, για παράδειγμα. Και εδώ είναι σημαντικό ο, ο κλάδος αυτός. Για... Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την προστασία των ποταμών, σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες ε, των ε, ποταμών και τις ζημιές που προκαλούνται. Άρα εμείς μαζί με τα κρατημέλη, μαζί με τις περιοχές και τις κοινότητες θα πρέπει να δούμε ακριβώς που χρειάζονται επενδύσεις προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας και νομίζω ότι έχουμε μέσα κοιτάτε τι γίνεται με τα ποσοστά απορρόφησης και ας περάσουμε λοιπόν και αυτό το μέσο. Ευκρινιστική. Κοιτάξτε. Λοιπόν, είμαι από τη Ρουμανία και είμαι ικανοποιημένη που γνωρίζετε την πραγματικότητα στη χώρα μου. Όπως γνωρίζετε, ήδη ήσασταν επίτροπος δύο φορές Στη χώρα μου, τη Ρουμανία, δεν είχαμε τη δυνατότητα να απορροφήσουμε τα ευρωπαϊκού πόρου για τι βασικέ υποδομέ. Κάποια προγράμματα πέτυχαν, κάποια άλλα όχι. Και πώ θα μπορούσαμε να δεσμευτούμε, να εφαρμόσουμε πιο περίπλοκα περιβαλλοντικά προγράμματα αν δεν αλλάξει όλη η στρατηγική. Αν η στρατηγική δεν αλλάξει, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Χωρί υποδομέ βασικέ, χωρίς πράσινες υποδομές βασικές. Είσαστε έτοιμοι να αλλάξετε λοιπόν στρατηγική, έτοιμος να αλλάξετε στρατηγική. Also, weder kann noch will Ούτε μπορώ, ούτε θέλω να κάνω τη δουλειά της Μελλοντικής Επιτρόπου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αλλά, ως μέλος του Σώματος των ε, Επιτρόπων και ως πρώην Επιτρόπος Περιφέρειας και αν επιβεβαιώσετε και ως Επίτροπος Προϋπολογισμού, αυτό που μπορώ να κάνω και αυτό που προσπαθώ να κάνω και να μεταφέρω ως μήνυμα τα τελευταίες δύο ώρες είναι το εξής. Στην εφαρμογή της, ε, στην υλοποίηση των πολιτικών μας στόχων ως Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσουμε η υλοποίηση της πολιτικής να ανταποκρίνεται στην εξαγγελία των στόχων. Κάποιες χώρες και η Ρουμανία είναι μία από αυτές. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να τις ε, βοηθούμε προκειμένου να αυξήσουν το ποσοστό απορρόφησης προκειμένου να, να αξιοποιήσουν τελικά τους πόρους τους οποίους τους διαθέτουμε. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι υπάρχουν τα χρήματα, δυστυχώς όμως δεν χρησιμοποιούνται. Θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν σωστός προγραμματισμός για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Και τώρα, ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ελέγχου Προϋπολογισμού, θα αναλάβω την Προεδρία και θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον Γιώχαν Φαν Όφερτφέλντε. Γι' αυτό και ανέλαβε την Προεδρία. Κύριε Επίτροπε, Ας θεωρήσουμε το εξή σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι το Συμβούλιο δεν καταλήγει σε συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις, ε, τους ίδιους πόρους ε, του χρόνου. Και ας υποθέσουμε επίσης ότι το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, αν συμφωνηθεί, είναι πολύ πιο χαμηλά από τη δικιά σας πρόταση. Θα υπάρξουν περικοπές, η πρόταση βέβαια της Νέας Προέδρου θα είναι εν μέρη μέσα, αλλά θα υπάρχουν επιπλέον περικοπές και τέλος δεν θα έχουμε νέους ίδιους σπόρους. Αυτό είναι το σενάριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βέβαια δεν επιτυχάνεται έτσι ο στόχος ούτε της προηγούμενης ούτε της μελλοντική επιτροπής. Εσείς λοιπόν τι θα κάνετε με το Συμβούλιο για να θα προσπαθήσετε να μας πείσετε ότι αυτό είναι και δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα παραπάνω ή θα πάτε στο Συμβούλιο και θα πιέσετε ε, προσπαθώντας να πετύχετε εκεί εκ νέου διαπραγματεύσεις ή θα πιέσετε το Κοινοβούλιο και τελικά εμάς θα κατηγορήσετε στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε να έχουμε συμφωνία μέχρι το τέλος ψυχολογικούς όρους θα έλεγα ότι πρόκειται για... Προσπαθείτε να εκμεύσετε πληροφορίες. Όπως ξέρετε είμαι μέλος ε, όχι μόνο μια πολιτική ομάδα, αλλά μιας πολιτική ομάδα που βλέπει τα πάντα ε, μισογεμάτα, όχι μισοάδια. Γι' αυτό θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και δεν πρόκειται να κάνω πίσω ούτε στην ε, κοινή γνώμη και θα πάω λοιπόν στα κάτι μελη και θα παρουσιαστώ στη δημοσιότητα και θα προκαλέσω αναστάτωση και σουσουρό σε ό,τι αφορά τις χώρες που κάνουν πίσω για να ξεκαθαρίσω τι είναι το διακύβευμα εδώ. Γιατί θεωρώ ότι όλη η Ευρώπη και όλος ε, ο πληθυσμός πρέπει και αισθάνεται μια μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις στον τομέα του κλίματος, επενδύσεις σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεις σε μια ανταγωνιστική μελλοντική οικονομία. Ο κόσμος θέλει επενδύσεις λοιπόν στην ε, έρευνα για μέσα τα οποία χρειάζονται για την υποστήριξη των νεοφιών επιχειρήσεων. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα πετύχουμε με πιο λίγους πόρους. Είναι απλό. Εδώ λοιπόν είμαστε σύμμαχοι και δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Θεωρώ ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρξει συμφωνία κάτω από το επίπεδο των όσων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσουμε δηλαδή τους στόχους μας. Θα είναι δύσκολες οι πολιτικές συζητήσεις, αλλά αν δράσουμε μαζί και αν συνεργαστούμε, θεωρώ ότι θα είναι μισογεμάτο, μη σας πω και σχεδόν γεμάτο το ποτήρι. you. like Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δείξω και ένα άλλο ζήτημα τώρα και να συνδέσω κάπως τη, τα προηγούμενα καθήκοντά σας και τα επόμενα εφόσον επιβεβαιωθείτε βέβαια στη θέση αυτή. Έχετε ασχοληθεί πολύ με τα σύνορα της Ευρώπης, με το μεταναστευτικό, με τη στρατηγική για τα Βαλκάνια και δεδομένου ότι και η Επιτροπή μας ασχολείται πολύ με γεωπολιτικά ζητήματα σε σχέση με το έργο μας, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα με το σημερινό προϋπολογισμό, πώς θα καταφέρουμε να φέρουμε σε πέρες τις φιλοδοξίες μας για τη θέση μας ε, στο, στην γεωπολιτική σκηνή και για τις σχέσεις μας με τις γείτονες χώρες. Κοιτάξτε, δεν θέλω νέα ακρόαση, έτσι δεν το πάω να με ξανακαλέσετε εδώ. Πάντως πολλά θα μπορούσε να πει κανείς εδώ. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αύξηση για όλον αυτό τον προπολογισμό τη τάξη του 24% αν δεν απατώμε, με τρεις παρεμβάσεις, ε, Δυτικά Βαλκάνια είναι το ένα, διεύρυνση, προένταξη, γειτονία και Αφρική. Και ακριβώς σε αυτούς τους τομείς εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ακριβώς γι' αυτό και οι χώρες που είναι πιο πρόθυμες πρέπει να πιστούν, πρέπει να τους εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό να επενδύουμε στην Αφρική. Ε, πάντα λέω εγώ ότι η προστασία των εξωτερικών μας συνόρων ξεκινάει όχι στα εξωτερικά μας σύνορα, ξεκινάει πολύ πιο μακριά. Πρέπει πρώτα να βοηθήσουμε την κάθε αφρικανική χώρα να αντιστέκεται καλύτερα. Πέρασε το λεπτό μου και πάλι θα μπορούσα να σας πω πολλά από την εμπειρία που έχω σε αυτό το τομέα. Πάντως έχουμε ξεκινήσει, έχουν ήδη γίνει πολλά και ελπίζω ότι θα συνεχιστούν οι επιτυχίες μας. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να περάσουμε στους ε, ομιλητές από την Επιτροπή Ελέγχων του Προπολογισμού, κύριο Στεχόφσκι. Αγαπητέ Επίτροπε, μια ερώτηση έχω θα ξεκινήσω με γενικό σχόλιο. Όποιος δεν ήταν στην Επιτροπή Προπολογισμών, ποτέ δεν ξέρει τι σημαίνει κόλαση. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και στις ακροάσεις μας. Νομίζω ότι αυτό το ψήσιμο θα σας δείξει ότι οι ερωτήσεις μας δεν είναι πολύ εύκολες. Σας έχουμε ψήσει. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίες της ξεκίνησαν διάφορες έρευνες όσον αφορά πάτε, όσον αφορά τα οικονομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλυση συγκρούσεων συμφερόντων έκαναν. Και αυτό ε, οδήγησε σε διοικητικές δράσεις και νομικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο που πιθανότατα δεν θα ανελάμβανονται διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του το τρόπος έχει ελέγξει ανεξάρτητα το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτηση. Πόσο οικονομικούς και προσωπικούς πόρους θα αφιερώσετε για έλεγχο και έρευνα όσον αφορά την κατάχρηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη, τα στοιχεία που δίνουν οι αρχές των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων δεν είναι πάντα αξιόπιστα. Συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πει να τα στοιχεία. Σχεδιάζεται να ενισχύσετε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, είχα τη χαρά τελευταία δεκαετία να είμαι στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού ε, πολλέ φορέ. Όχι στην Επιτροπή Προπολογισμών, στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Και πολύ χαίρομαι να συνεχίσουμε. Όπω ήδη ανέφερα, έχουμε πάνω από 500 άτομα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που ασχολούνται με ελέγχου. 385 στην Όλαφ. Έχουμε ανθρώπους στη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Στις υπηρεσίες για τη μάχη περίπου 400 Είμαστε αρκετά επιτυχείς όσον αφορά τον εντοπισμό ατασταλιών. Δράτω με τη ευκαιρία όμως για να πω ότι πάντα μιλάμε πολύ για το ποσοστό σφάλματος και πολλοί συγχαίουν το σφάλμα με την απάτη. Και δόξα το Θεό, το ποσοστό απάτης μέσα στα σφάλματα είναι λιγότερο από 1% αλλά και πάλι είναι ψηλό. Μηδέν θα ήταν το ιδανικό. Είναι σημαντικό όμως να κάνω τη διάκριση μεταξύ σφάλματος και απάτης. Ακόμα και αν υπάρχει σφάλμα, πρέπει να γίνουν οικονομικές διορθώσεις. Ένας από τους λόγους για τον οποίο έχουμε ακόμα σφάλματα και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος σφαλμάτων, είναι ότι καμιά φορά οι κανονισμοί μας είναι πολύ περίπλοκη, δυσκολότατη. Και ένα μεγάλο ζήτημα είναι το πώς θα πλουστεύσουμε αυτούς. Και αυτή η έννοια της απλούστευσης με συνοδεύει από όταν ήρθα εδώ. Αυτή τη φορά στην πολιτική συνοχής προτάθηκαν 80 απλουστεύσεις. Τώρα από τον τριμερή διάλογο και τις διαπραγματεύσεις εξαρτάται πόσες από αυτές θα εφαρμοστούν. Κατά αποκοπήν ποσά, φερρυπίν, επιλεξιμότητα, ΦΠΑ. Στόχος η μείωση του κινδύνου σφαλμάτων. Και εξ αυτού προλαμβάνουμε το ότι οι τελικοί δικαιούχοι να έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και βασίζομαι σε εσά και στις τριμερεί στους διαλόγους να δεχτείτε αυτή την έννοια της απλούστευσης. Διευκρινιστική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Η δεύτερη μου ερώτηση σχετίζεται με την Όλαφ. Είναι φορέας που έχει τη φήμη ότι έχει πλήρη ανεξάρτητο ερευνητή για τις απάτσες της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Θα εξακολουθεί να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της η Όλαφ αν οι ερευνητέ, οι ελεγκτές της μεταφραστούν στο EPPO που θα έχει διαφορετικό καθήκον. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και δεύτερον, η σύγκρουση συμφερόντων. Ε, επίτροπε, υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν μεγάλα προβλήματα με τη σύγκρουση ε, συμφερόντων σε πολιτικούς υψηλού επίπεδου. Τι θα κάνετε γι' αυτό. και πώς θα βοηθήσετε πολλές αρχές σε πολλές χώρες που έχουν αυτό το πρόβλημα. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ένα λεπτό. Όσον αφορά το προσωπικό της Όλαφ και της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. πρέπει να συνεργαστούν. Θα συνεργαστούν. Αναφέρεστε σε συμφωνία της κυρίας Γιώργεβα με τον κύριο Άσλμπορν από το παρελθόν για μεταφορά προσωπικού, μετακίνηση προσωπικού. 2015-2016 νομίζω τη συνήθη. Βασιζόταν σε πρώτες Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έγινε τότε όσον αφορά τη δομή της μελλοντική Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Εν τω μεταξύ έχουν περάσει οι κανονισμοί. Λόγω των διαπραγματεύσεων ο χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Αγγελία έχει κάπω αλλάξει. Οπότε οι ανάγκε από πλευρά προσωπικού πρέπει να προσαρμοστούν δεόντως. Αυτό έγινε και τώρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ξεκινήσει τη λειτουργία της και μετά θα δούμε ποιες θα είναι οι συμπληρωματικές ανάγκες. Αλλά η Όλαφ εν γέννη είναι σημαντικότατος φορέας για λόγους ε, ελεγκτικούς και ερευνητικούς και στο μέλλον ε, το, το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού της Όλαφ θα παραμείνει στις Βρυξέλλες, στην τριπτική πλειοψηφία, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν έχω χρόνο να απαντήσω. Εν συντομία, Αναφερθήκατε σε ιδιαίτερη ειδική περίπτωση, ξέρουμε τι εννοείται. Οικονομική ζημία για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εκεί σταματήσαμε τις πληρωμές και συμφωνήσαμε στις τσεχικές αρχές να μην υποβάλουν τιμολόγια. Απ' την άλλη σταματήσαμε δηλαδή τη διαδικασία. Συνεχίζονται οι έλεγχοι. Περιφαίνουμε το Δεκέμβριο για τη Ρίτζο και άγρι τον Ιανουάριο και όταν έχουμε τα πορίσματα των ερευνών θα επανέλθουμε και σας ενημερώσω σχετικά με αυτά. Ευχαριστώ. Ο Κλάις Μέντα, συντονιστής της ε, Σοσιαλιστικών και Δημοκρατών στο... στην ΚΟΝΤ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Οριστέντα, Επίτροπε, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το κράτος δικαίου αποτελεί πλήρως μέρος του νέου προπολογισμού και ο τριμερής διάλογος για αυτό το μηχανισμό πρέπει να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα στηρίξετε επίσης την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προστατεύσει τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών ε, ταμείων να φροντίσετε να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και επίση συμφωνείτε ότι πρέπει να είναι πολύ λεπτομερής ο ρόλος του Κοινοβουλίου όταν μιλάμε για αυτό τον μηχανισμό κράτους δικαίου. Έχουμε μια πρόταση επιτάπητος σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και την εφαρμογή του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά τη χρήση ευρωπαϊκών ε, πόρων. Και θεωρώ ότι είναι σωστή και λογική πρόταση. Τι λέει ουσιαστικά αυτή η πρόταση όταν πρόκειται για ευρωπαϊκούς πόρους, η σωστή χρήση των πόρων και σε ό,τι αφορά ε, κρατικούς πόρους, μίλησα για το ΦΠΑ προηγουμένως, όταν ε, δεν υπάρχει τέτοια εγγύηση και υπάρχουν ε, ελλείμματα σε κάποια χώρα, στο μέλλον ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε. Αυτό που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, αυτό είναι το τμήμα της πρότασης άλλωστε, είναι τελικά να μην πλήττεται ο τελικός δικαιούχος. Αν υπάρξει αναστολή των πληρωμών μας, προς, μια, προς ένα κράτος, κράτος μέλος, το κράτος μέλος υποχρεούται, εφόσον έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, να υποβάλει τις πληρωμές προς τον τελικό δικαιούχο. Αυτό προτείνεται ως διαδικασία. Συμπληρωματική ερώτηση. Μπορείτε να μας εγγυθεί ότι ο μηχανισμός αυτός σχετικά με το κράτος δικαίου θα εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο εξίσου σε όλες τις χώρες. Δηλαδή ό,τι επιτρέπεται σε κάποιες χώρες πρέπει να επιτρέπεται σε όλες τις χώρες και ό,τι απαγορεύουμε σε κάποιες χώρες πρέπει να απαγορεύεται σε όλες τις χώρες μέλη. Μας το αυτό. Απόλυτα. Και νομίζω ότι εδώ αυτό που είναι πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο είναι το εξή. Τον Ιούνιο Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθο, αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον ετησίω να γίνεται μια αξιολόγηση κράτους δικαίου για όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό βάσει κοινών διαδικασιών και κανόνων, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα και να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι κάποιοι αντιμετωπίζονται με χειρότερο ή με καλύτερο τρόπο. Ω Επίτροπο Περιφερειακή Ανάπτυξη ε, με τον τότε συναδελφό μου, τον Όλι Ρεν, εργάστηκα προς την κατεύθυνση αυτή και σε μια χώρα που δεν μπορούσαμε να εγγυηθούμε την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας απειλήσαμε με την αναστολή των ε, πληρωμών. Υπήρχε η νομική αυτή δυνατότητα, κινητοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά τότε και γι' αυτό λοιπόν αναπτύξαμε ένα τύπο μαθηματικό για το πώς θα υπολογίσουμε ε, την αναστολή των πόρων αυτών, τι ποσό θα ανασταλεί, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει εντύπωση ασφαλμένα ότι κάποιες χώρες ε, έχουν καλύτερη μεταχείριση ή όχι αναφέρατε τη λέξη κλειδί, ίση αντιμετώπιση των χωρών ανεξάρτητα από το αν είναι μικρές ή μεγάλες. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Επόμενη ερώτηση. Η κυρία η κυρια φοβινιο Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαρβαμά πήρε το λόγο. Διακόπτη, Πρόεδρος. Η Καταλήν ξέρει, είπα, ότι έχει το λόγο. Λυπούμε, λέει ο κύριο Σαρβαμά. Παρακαλώ, εσείς. Σας ευχαριστώ. Θέλω να επικεντρωθώ στην απλοποίηση. Γιατί όσο χρόνο μπορώ, συναντάω τους ε, εκλογείς μου και τι ακούω από αυτού, ότι έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία, ότι κρατάει πάρα πολύ χρόνο το να βρούνε πληροφορίες και μπερδεύονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, κάτι το οποίο δυσκολεύει την πρόσβαση στο Ταμείο Συνοχής. Και αυτό ισχύει κυρίω για ανθρώπους που ζουν στην Ήπεθρο, σε ορεινέ περιοχές ή αυτού που έχουν περισσότερε δυσκολίε για διάφορου λόγους. Οπότε, δεν θα έπρεπε να γίνονται πιο εύκολες ε, οι διαδικασίες για την πληρωμή ενισχύσεων. Θα πρέπει να μπορούν να καταλαβαίνουν δικαιώχοι τι συμβαίνει. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν πιο αποτελεσματικά να αξιολογήσουμε αυτές τις διαδικασίες ώστε να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση, η προσβασιμότητα στα κονδύλια, να καταλαβαίνει ο κόσμος επίσης καλύτερα. Εσείς λοιπόν, τι θα κάνετε για την απλοποίηση και τι νέα εργαλεία θα στη διαδικασία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε πολλές χώρες όπου σε κάποιες χώρες ακόμα και οι κυβερνήσεις λένε ότι δεν θέλουμε διαφορετικά ταμεία γιατί είναι τόσο περίπλοκα που τι να τα κάνουμε. Και σε κάποιους τομείς υπάρχουν και επιχειρήσεις ε, που δηλώνουν ότι είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Έχουμε δύο δυνατότητες ε, αντιμετώπισης, αλληλοσυνδεόμενε. Η μία είναι η εξή. από πλευράς μα να κάνουμε ε, απλουστεύσει, και είπα ότι στον τομέα των ε, περιφερειακών ταμείων έχουμε περίπου 80 μονομένα μέτρα τα οποία προτείναμε για την επόμενη ε, περίοδο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και ελπίζω να επιβιώσουν και οι 80 αυτές προτάσεις από τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τα μέσα τα οποία μπορούν να κινητοποιηθούν. Και κάτι άλλο, το δεύτερο. Μπορούμε σε όλα τα κράτη-μέλη να υπάρχει μια τάση που ονομάζεται golden plating. Δηλαδή, να επιβάλλουμε άλλη μια, ένα άλλο επίπεδο ελέγχων για να κάνουμε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Και τα δύο λοιπόν θα πρέπει να τα εξετάσουμε και τα δύο θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των μέσων για τους τελικούς ε, δικαιούχους. Ε. Μία δυνατότητα ε, λοιπόν, που αναφέρθηκε ήταν τα ποσά κατά αποκοπή, λάμψαμς, προκειμένου να μην πρέπει να παρουσιάσετε κάθε μικρολεπτομέρεια. Να Δίνουμε δυνατότητα προώθησης μέχρι 5 εκατομμύρια προκειμένου να απλοποιήσουμε την κατάσταση και να μειώσουμε και τον κίνδυνο τα ασταλείων. Ευχαριστώ πολύ. πληρωματική ερώτηση τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτροπε και τώρα έχουμε τον κύριο Σαρβαμά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από τον αγαπητό συνάδελφο, από την κυρία Σέχ. Στα 8 χρόνια μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Προπολογισμών συνήθισα να λειτουργούν σαν ελβετικό ρολόι τα θέματα προπολογισμού. Εξέτασα μόνο τον κατάλογο των επισήμων ομιλητών κυρία, απουσίαζε μια κυρία και εγώ νόμιζα ότι θα, θα πάρω εγώ τη θέση, γι' αυτό πήρα το λόγο, ζητώ συγγνώμη. Μου κλέψαν και την ερώτηση. Παρόλο που πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και το κάτω δικαίου ετέθη τρει φορές ή τέσσερι φορές, θα ρωτήσω λοιπόν το εξή. μετά από αυτά που είπε ο πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών, που έκανε μια ερώτηση, ήταν σημαντικότατη ερώτηση, δεν νομίζω ότι πήρε την απάντηση που μας αξίζει. Δηλαδή, παρόλο που δεν θεωρείται ότι είναι δυνατόν το τελικό αποτέλεσμα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου να είναι χαμηλότερο ποσό από αυτό της προτάσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πάντως δυνατόν το τελικό αποτέλεσμα να είναι πολύ κοντά ή να είναι το ίδιο. Θέλω συγκεκριμένη απάντηση. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εσά σαν έντιμος διαμεσολαβητής σε αυτή την κατάσταση, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις και τα καθήκοντα που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τίποτα λιγότερο από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήδη είναι πολύ μικρό ποσό. Ευχαριστώ. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ και να περιμένετε είναι ότι θα τους επόμενους δύο μήνες θα αναλώσω το χρόνο μου, σχεδόν όλο μου το χρόνο, αλλά έχω και άλλες ευθύνες, όχι μόνο για να διαπραγματευτώ στις Βρυξέλλες μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Προεδρίας του Συμβουλίου, αλλά να πάω και στα κράτη-μέλη να μιλήσω όχι μόνο με τους αξιωματούχους, να απευθυνθώ στο λαό, στο κοινό. Να ζητήσω ε, υποστήριξη του λαού για τους κοινούς μας στόχους. Δεν μπορώ να εγγυηθώ συγκεκριμένο αποτέλεσμα όσον αφορά ποσοστά και ποσό. Θα κάνω όμως ό,τι μπορώ, ούτω ώστε τουλάχιστον να φτάσουμε στο επίπεδο της πρότασης της παρούσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το ελάχιστο. Πέραν αυτού δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι και θέμα άλλων ζητημάτων που αναφέρεται. Ιδίους πόρους, ε, να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε το επίπεδο της ευελιξίας, να ε, εισαχθεί το θέμα του κράτους δικαίου, αφορά όλα αυτά και εξυγχρονισμό της πολιτικής για να μπορούμε να πουλήσουμε αυτές τις αρχές στους πολίτες. Βασικό θέμα είναι να στραφούμε στους πολίτες, να εξηγήσουμε γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα. Ο Έτιγκερ λέει ότι όταν παράγεις 100 ευρώ, λέει, πρέπει να πληρώνεις 50 ευρώ στη χώρα. Και 49 ευρώ μένουν στον εθνικό προπολογισμό και ένα ευρώ μόνο πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες τις πολιτικές που χρειάζονται και ζητούν οι πολίτες μας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και σίγουρα αυτό θα κάνω. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα τμήμα του να είναι κανείς ένας έντιμος διαμεσολαβητής, να λέει στον κόσμο περί πρόκειται, ποιο είναι το διακύβευμα, τι γίνεται άμα δεν έχουμε παρκή χρήματα. Διότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός με αυτό το 1% κατευθύνει τις πολιτικές όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης, αλλά επίσης εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές στα κράτη-μέλη. Κάθε προσπάθεια χρειάζεται για να πάρουμε και άλλα χρήματα. Δεν θα ήταν σοβαρό τώρα να σας δώσω κάποια υπόσχεση για συγκεκριμένο ποσοστό. Μπορώ μόνο να υποσχεθώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ και δεν θα σταματήσω πριν πετύχω τουλάχιστον τα αναγκαία. Διευκρινιστική ερώτηση. Σύντομα παρακαλώ, διότι οι πρώτες ερωτήσεις ε, ξεπεράσανε το, το χρόνο κατά ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σχετίζεται με την πρώτη μου ερώτηση αυτή. Υπόσχεστε ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού του Κοινοβουλίου ότι θα εξετάσετε προσεκτικά τις ανάγκες της Όλαφ και να λάβετε υπόψη την ερευνητική εμπειρία που έχουν για να παραμείνουν σε αυτή την πόλη και να μην φύγει Όλαφ και να πάει στο Λουξεμβούργο. Απάντηση για να εξοικονομήσουμε χρόνο, θα απάντησή μου θα είναι ναι. Μα φανταστική, τέλεια απάντηση κύριε Επιτροπέ με το επιθυμητό περιεχόμενο κιόλα. Η Ιζαμπέλ Καρσία Μούνιο είναι η επόμενη. Από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Χάν, εδώ βρίσκομαι. Μια από τι κύριε αποστολέ και καθήκοντα του νέου Επιτρόπου θα είναι να ελέγχει ακριβώ το έργο της Επιτροπής στον έλεγχο των συμφερόντων των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάσαμε στις απαντήσεις σας ότι θα ενημερώνετε την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών για τις ε, εισπράκτης, την ανάκτηση χρημάτων δηλαδή που έχει πετύχει Όλαφ. Μπορείτε όμως να μας πείτε πώς θα ενισχύσετε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστατεύει οικονομικά σφαίροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες. Επίσης, οι σοσιαλδημοκράτες ανησυχούν για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής εισαγγελία, γιατί αυτό σημαίνει ότι ίσως η Όλαφ να μπορεί να κάνει λιγότερα πράγματα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και ο πυρήνας των αρμοδιοτήτων της. Εσείς τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό τη στιγμή που δεν έχει πετύχει ακόμα πλήρως τον ε, στόχο της η υπηρεσία της όλα. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας πρώτα απ' όλα. Πάντως, αν μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι ε, με το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη. Ελπίζω να συμμετέχουν και άλλες, όπως η Σουηδία, η Δανία. Και αυτό να οδηγήσει και τις υπόλοιπες να συμμετέχουν. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, ήδη με την Όλαφ προστατεύουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ένα βήμα προς τα μπρος, γιατί πρόκειται για διασυνοριακή συνεργασία. Είναι καλό να την έχουμε. Δεν είναι ακόμα τέλεια, αλλά είναι σημαντικό να αρχίσουν να λειτουργούν. 1η Ιανουαρίου του 2020 θα γίνει αυτό. Και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο κύριος Ρέιντερς, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι συναδερφός μου στο μέλλον, πέρασε την χτεσίνη ακρόση και θα συνεργαστώ μαζί του. Συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Ωραία. Είπατε ότι δεν μπορείτε να δεχτείτε να υπάρχουν χώρες που είναι εκτός. Εσείς τι μέτρα θα πάρετε ώστε να πείσετε τις χώρες αυτές να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επαναλαμβάνω και την δεύτερη ερώτησή μου που δεν απαντήθηκε και ήταν για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Δεν νομίζετε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής εισαγγελία όσο δεν έχει φανεί ότι είναι σε θέση να λειτουργήσει ικανοποιητικά και πραγματικά να προστατεύσει τα ε, οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης. Το δεύτερο μέρος δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μια συγκεκριμένη αποστολή τώρα, έτσι. Και υπάρχουν ιδέες η πρόεδρος της Επιτροπής έχει προτείνει και ο Ντιδιέ Ρέιντες χθες ήταν ξεκάθαρος γιατί είπε ας αρχίσουμε με τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής εισαγγελία, να δούμε πώς θα λειτουργήσει και μετά αν τα πράγματα πάνε καλά, αν είναι αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αν υπάρχει ανάγκη επέκτασης των αρμοδιοτήτων, ώστε να προσθεθούν και άλλα καθήκοντα, τότε δεν θα διστάσουμε να τροποποιήσουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τώρα για το πώς θα πείσουμε ε, τις χώρες που δεν συμμετέχουν ήδη, δεν μπορούμε να τις αναγκάσουμε, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα χάσω καμία ευκαιρία προκειμένου να ε, προσπαθήσω να τις πείσω. Είναι και θέμα ε, φήμης βλέπετε για τις χώρες που δεν συμμετέχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νομίζω ότι δεν είναι καν προς το δικό τους το συμφέρον να μείνουν εκτός. Σε ευχαριστώ πολύ και τώρα να ακούσουμε του πράσινους, τον Μίκουλα Πέξα. Αγαπητέ Επίτροπε, Κατάρχά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε εδώ στην Επιτροπή μα, στις Επιτροπές μας για να απαντήσετε στι ερωτήσει μα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Η τριμερή συμφωνία που έχει υπογραφεί από την Επιτροπή το αμα, Συνέδριο θα εκπνεύσει το 2020 σε ό,τι αφορά τις ε, δραστηριότητες που παρακολουθεί η τράπεζα και σε ό,τι αφορά το γενικό προπολογισμό. Ω Επίτροπος θα εξασφαλίσετε ότι τα υφιστάμενα εμπόδια σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη τριμερή συμφωνία θα αφαιρεθούν και το Ευρωπαϊκό Ελεκτρικό Συνέδριο θα μπορεί να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς τους Ευρωπαίους πολίτες τι γίνεται σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα και την διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δέωση επιμέλεια των ευρωπαϊκών επενδύσεων και τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα, τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κύριε Επιτροπέ, καταλαβαίνω την ερώτησή σας και ως προς το περιεχόμενό της δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ανεξάρτητο σώμα και διέπεται από ξεχωριστούς κανονισμούς. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του. Είναι απόφαση των κρατών μελών. το τι πιστεύουν ότι είναι χρήσιμο σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και κατά πόσον το λεκτικό συνέδριο θα πρέπει να ελέγχει την ΕΤΕΠ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να έχω μια δημόσια τουλάχιστον άποψη από αυτού. Κάτι άλλο για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω ωστόσο. Αν η ΕΤΕΠ χρησιμοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους για κάποια προγράμματα, το ελεκτικό συνέδριο έχει δυνατότητα να ελέγξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Ε, περαιτέρω ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, απάντηση τουλάχιστον υπό τη μορφή αυτή. Η ΕΤΕΠ ε, αλλάζει στην παρούσα φάση την πολιτική της και λαμβάνει, μάλλον δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις δαπάνες για την αλλαγή του κλίματος. Ως επίτροπος, τι εννοείται με επενδύσεις για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. τι μπορεί να χρηματοδοτεί από την, με την πολιτική της αυτή η ΕΤΕΠ. Ο Επιτροπός. Κοιτάξτε. Είναι πολύ πιθανόν η ΕΤΕΠ να συμμετέχει στο Ταμείο Δικής Μετάβασης με τα οικονομικά της μέσα. Και αυτό είναι το ένα στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο θα μπορούσε να είναι το εξής. Να, μη δίδονται προϊόντα πιστώσεις για την οικοδόμηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας με άνθρακα, με λιχνίτη. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδέα. Υπάρχουν τρόποι για να καθοριστεί το πού μπορούν να γίνουν επενδύσει και πού όχι. Και φαντάζομαι ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει στου κόλπου τη ΕΤΕΠ και μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για να δούμε πώ θα υπάρξει αυτή η μετάβαση για να γίνει μια πράσινη τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωση και πώς θα επαναπροσδιοριστεί η εταιρική πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτροπε. Ματέο Αντινόλφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, όπως ποτέ, πρέπει να επιλέξει κρίσιμες πολιτικές που αναπόφευκτα θα αντικατοπτριστούν στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να καταλάβουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον προτίθεται να γίνει σπίτι των εθνικών, των εθνών της των ευρωπαϊκών κρατών, σεβόμενη την κυριαρχία των κρατών εθνών, ή να είναι μια λέσχη που αυτοπροσδιορίζεται, που θέλει να αντικαταστήσει τα διάφορα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών μελών. Όταν συζητάμε την ενίσχυση του κράτους δικαίου για τους πολίτες να έχουμε και έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών ενώ οι φορολογουμένοι πλητών την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Εξωτερική Δράση που επαναλαμβάνει υπηρεσίε εθνικές και σας ρωτώ μετά από αυτά πώς προτίθεστε να εγγυηθείτε μια υγιή αναθεώρηση των σπαταλών και πραγματική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας υπάρχουν εκατομμύρια επικατομμυρίων Ευρωπαίοι πολίτες που ζητούν δυνατά να προσέξουμε τι δαπάνε του προπολογισμού και να εξετάσουμε αν υπάρχουν ατασταλίε. Τι απαντάτε σε αυτού του πολίτε οι οποίοι ε, έχουν αυτό το πρόβλημα και διαμαρτύρονται γι' αυτό. Σα ευχαριστώ. Ε, ε, τι να απαντήσω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τους εκλεγμένους εκπροσώπους, τους βουλευτές που έχουν καθήκον και ρόλο σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Αυτό είναι αυτονόητο δικαίωμα του Κοινοβουλίου. Από την άλλη, ορθώς επισημάνατε και την ε, αρχή επικουρικότητας. Η αρχή επικουρικότητας κατοχυρώνεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποδυναμώσει κανείς ή να αναιρέσει την αρχή της επικουρικότητας. Είμαστε τμήματα της Ευρώπης και πάντα αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να γίνει η κάθε δουλειά. Αυτή η συζήτηση λοιπόν είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνεται διαρκώς και σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του επόμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να συζητήσουμε ποια είναι τα καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν σε περιφερειακό, κρατικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και σε δημοσιονομικά μέτρα. Η δική σας ε, λοιπόν ευθύνη είναι να συμμετέχετε στη συζήτηση αυτή και να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή υπεραξία και ότι παράλληλα θα τηρείται και η αρχή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Επίτροπε. Ένα follow-up ε, σύντομο όμως. Grazie. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, επανειλημμένα λέτε ότι προτίθεστε να ακούσετε τους πολίτες των διαφόρων κρατών μελών και να σταθείτε σε αυτούς. Οι συνάδελφοι της οι μελλοντικοί επίτροποι δεν λαμβάνουν υπόψη στην Ευρώπη. Οι πολίτες δοκιμάζονται σκληρά από τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται από την Τρόικα και αντιμετωπίζουν απόλυτη φτώχεια. Τι προτίθεστε να κάνετε. Μάλλον ε, ακόμα και μπορούν να φάνε στο φαγητό κάθε μέρα. Κύριε Επίτροπε, θέλουμε να τονίσουμε εκείνες τις δαπάνες που από χρόνια έχουν γίνει μόνο οικονομικά μη βιώσιμες αυτές οι δαπάνες και σπατάλες, αλλά ηθικά παράδεκτες. Όπως το κόστος που όσον αφορά τις του Κοινοβουλίου, Βρυξέλλες, Στρασβούργο και Λουξεμβούργο, το Κοινοβούλιο έχει τι έδρες. Και το κόστος του υπερβολικό οργάνων όπως είναι τα χρήματα που δίνονται τα προταξιακά στην Τουρκία και πολλά άλλα χρήματα. Πότε θα σταματήσουν αυτές οι σπατάλες και πώς θα είσαστε πιο κοντά στις ανάγκες και τις απαιτήσει των πολιτών. Επιτροπός, ε, αυτή είναι η ουσία της Ευρώπης. Το ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στον ίδιο κορφανά, εδώ στις Βρυξέλλες. ότι είμαστε παρόντας σε όλη την Ευρώπη. Και ο κόσμο σε πολλέ περιπτώσει λέει: Μα αυτή εκείνη τη αυτοί αυτή εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε και ποιου εκπροσωπούμε. Αν δεν είμαστε μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν είμαστε δήμαρχοι στην ε, χώρα μας ε, και αυτοί και οι δήμαρχοι είναι εκπρόσωποι μια κοινή Ευρώπη. Θα ήταν λοιπόν σφάλμα να κάνουμε τέτοια διαφοροποίηση και γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικό. Να τονίζουμε και στα γραφεία μας και παντού ότι αυτή η Ευρώπη ε, βρίσκεται παντού. Δεν εκτελήσεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Και το γεγονός ότι εσείς μου μιλάτε στα Ιταλικά εγώ σα απαντάω στα γερμανικά και ο κόσμο που μας ακούει στη μητρική του γλώσσα και αυτό αποτελεί ε, ένα αποτέλεσμα τη Ευρώπη που μα δείξει, μας δείχνει τι αξία υπάρχει. Και την ε, ποικιλομορφία της Ευρώπης, ε, την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι όλα αυτά κατοικοστίζουν. Γιατί σε τελική ανάλυση το κόστος αυτό μεταφράζεται στο ότι οι πολίτες ταυτίζονται τελικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές σε πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε συνδεθεί με υπηρεσίες, με οργανισμούς και όλοι αυτοί μας εκπροσωπούν. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά για να μην δημιουργηθεί εντύπωση ότι οι Βρυξέλλες, Ευρώπη είναι μόνο στις Βρυξέλλες. Όχι, παντού είναι Ευρώπη. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από την Επιτροπή Προπολογισμών, η κυρία Πρέτιε. Θα μιλήσω γαλλικά. Λέει κυρία Πελτιέ. Πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η διαμεσολαβήτρια ζήτησε να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες όσον αφορά τα υψηλά αξιώματα. Ότι χρειάζεται περισσότερη ισότητα στις ευκαιρίες, περισσότερη διαφάνεια. Οι προτάσεις του προκατόχου σας δεν είναι απαραίτητα ικανοποιητικέ από αυτού. Και όπω και εκείνο, έτσι και εσεί πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται καμία πραγματική αναθεώρηση. Μπορείτε λοιπόν να μα εξηγήσετε πώ μπορεί να αγνοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα του μοναδικού οργάνου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εκλέγεται δημοκρατικά και τις ε, συστάσεις επίσης της διαμεσολαβήτριας, δεν πιστεύετε ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι επιθυμητό και θα μπορούσε να βοηθήσει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαίους πολίτες. Παρακαλώ να απαντήσει ο επίτροπο. Νομίζω ότι η επιστολή του κυρίου Ότινγκερ προς την Πρόεδρο στα μέσα Αυγούστου αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τη μελλοντική διαμόρφωση της πολιτικής μας. Και φυσικά, βάσει αυτού, θα συνεχίσουμε τις εσωτερικές μας διαπραγματεύσεις. Εγώ είμαι πολύ υπέρ και αυτό ξεπερνάει το πλαίσιο. και σύντομα θα παρουσιάσω μια προσωπική, μια στρατηγική μάλλον για το προσωπικό για την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση που θα καλύπτει το θέμα αυτό πιο πολύ. Δεν το συζητήσαμε καθόλου σήμερα, αλλά υπάρχουν διάφορα που μπορούν να γίνουν και πρέπει να κάνουμε. Και εδώ λοιπόν θα κοιτάξουμε και το θέμα του διορισμού σε θέσεις διευθυντικές Εγώ είμαι σαφώς υπέρ για διάφορους λόγους όπου έχει νόημα να υπάρχουν ε, δημοσιοδιαγωνισμοί, αλλά να υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να δημιουργούμε, να αξιοποιούμε μάλλον ε, το άρθρο 7 του ιστορικού κανονισμού για να γίνονται μετακινήσεις, αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, διορισμών θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωση. Συμπληρωματική ερώτηση. Παρακαλώ. Με την απάντησή σας, εντάξει, φυσικά δεν φταίτε εσείς για τα όσα αποφάσισαν οι προκατοχοί σας. Εσείς, εγώ δεν ήμουν πριν ευρωβουλευτής, αλλά εσείς ήσασταν μέλος του Σώματος των Επιτρόπων. Οπότε, τι λέτε, η θέση σε ένα διοικητικό, σε μια διοικητική θέση αρκετά ε, υψηλή, δεν μπορεί να σοκάρει τους συμπολίτε μας. Ο νέος Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για παράδειγμα, επίσης διαμεσολαβήτρια, είπε ότι χρειαζόταν η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλεγε ότι αυτός ο ορισμός δεν ήταν σωστός. Ξεπέρναγε κάποια όρια. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Εσείς συμφωνείτε με το ΣΕΠ Μεσολαβήτρια και θα κάνετε κάτι ώστε τέτοιες καταστάσεις να μην επαναληφθούν όπως ήταν ο ορισμός αυτός του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δεν θέλω να επισέλθω σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας ε, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι όλα αυτά τα εξετάσατε ενδελεχώς εδώ στο Κοινοβούλιο. Να πω όμω ότι στο πλαίσιο των ε, κανονισμών και των ρυθμιστών συζητήθηκε το θέμα της ε, αξιοποίησης ε, των όρων αυτών σε ό,τι αφορά την πολιτική για το προσωπικό. Η αυτονομία του θεσμικών οργάνων ε, κατοχυρώνεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό καλούμε να το σεβαστώ. Αλλά σας ε, ομολογώ ότι εδώ πρόκειται για θέσεις οι οποίες ε, συγκεντρώνουν μεγάλη προσοχή από το κοινό εδώ στο στις Γι' αυτό λοιπόν και αυτό θα ληφθεί υπόψη στο μέλλον. Πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Θα προεδρεύσω οι τελευταίε δύο ερωτήσει που προέρχονται από τα μέλη τη Επιτροπή τη Νομική και ευχαριστώ του άλλου δύο προέδρου που με επιτρέπουν να το κάνω. Πρώτη ερώτηση από την Επιτροπή Γιούρη. Καρολίνε Στέλτερ από το ΕΛΚ. ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε ε, Επιτροπή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα θέματα κράτους δικαίου. Δεν θέλω να επαναλάβω ωστόσο ερωτήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι προσβλέπω σε μια εις συζήτηση του θέματος αυτό γιατί θεωρώ ότι το κράτο δικαίου αποτελεί βασικό τμήμα του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και υποθέτω ότι έχουμε την υποστήριξή σα Να αναφέρω ένα άλλο θέμα το οποίο και στο μέλλον θα μας απασχολήσει η ψηφιοποίηση, γιατί η πλήρης ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καθήκον σας. Γνωρίζετε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ότι κάθε άλλος εδώ και γι' αυτό θεωρώ ότι ήδη έχετε σχηματίσει μια εικόνα για το πόσο έχει προχωρήσει η ψηφιοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ. πώς αξιολογείτε την κατάσταση, τι τμήματα έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί αποτελεσματικά, υπάρχουν διάφορα άλλα τμήματα τα οποία εργάζονται με λογικό τρόπο, δεν το φαντάζομαι, και πώς θα διαθέσετε τους χρηματοοικονομικούς πόρους που χρειάζεται για την δημιουργία των ψηφιακών ικανοτήτων που χρειάζονται οι υπάλληλοι. Απάντηση. Κοιτάξτε, αποκλειστικά, αναλογικά δεν δουλεύει κανένας πλέον. Ε, το βάθος τώρα της ψηφιοποίησης μπορεί να διαφέρει. Εδώ, ναι, υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης σε κάθε περίπτωση. Συνολικά, όμως, έχουμε προχωρήσει. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Το πρόβλημα που επισημάνεται είναι ότι το σκηνικό είναι πολύ τερογενές σε ό,τι αφορά τα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται. Και βασικό λοιπόν καθήκον μας στο μέλλον θα είναι και μάλιστα η Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια ε, ήδη έχει ξεκινήσει τις εργασίες τη, δεν με περιμένει εμένα. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση. Αυτό και για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ε, της ε, γενικής, ε, μάλλον όχι για την ψηφιοποίηση των εργασιών της Επιτροπής, αλλά για την καλύτερη διαλειτουργικότητα, σε προκειμένου να είμαστε πιο γρήγοροι σε ό,τι αφορά την υποβολή αναφορών. Δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά ξέρω ότι απασχολεί διάφορο το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τη διαδικασία χορήγηση απαλλαγή. Πώ μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή. Αυτό εξαρτάται από διάφορου παράγοντε, αλλά μεταξύ άλλων εξαρτάται και από το κατά πόσον τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να χορηγήσουν τα δεδομένα που χρειάζονται γρήγορα. Και αυτό το κάνουν αν υπάρξει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα. Το Μάρτιο-Απρίλιο λοιπόν του ε, μεθεπόμενου έτους δεν θέλουμε να έχουμε Μάλλον δεν θέλουμε να έχουμε τη χορήγηση απαλλαγή 1,5 ε, χρόνο μετά. Το θέλουμε να το έχουμε ένα χρόνο μετά αν είναι πιο μεγάλη η ψηφιοποίηση και πιο καλή η αξιοποίηση των ικανότητων που έχουμε. Φαντάζομαι ότι οι βιντεοδιασκέψεις, για παράδειγμα, και αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Χρειάζονται χώροι ε, και στις Βρυξέλλες και αλλού. Εδώ όμως θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης πόρων αν έχουμε λιγότερες ανάγκες για έδρανα. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν έχουμε πιο πολλές ε, ψηφιακές δυνατότητες και οι οποίες να χρησιμοποιούνται για να υπάρχει επικοινωνία σε όλη την Ευρώπη. Ίσως ε, να μπορούμε να παρικόψουμε και κάποια ταξίδια. Ναι, Επίτροπε, έχετε ξεπεράσει το, το χρόνο που σας... Ε, δεν κοιτάξτε, είμαι τόσο ενθουσιώδης για το θέμα αυτό, δεν μπορώ να σταματήσω. Έχουμε όμως μια συλλογική ερώτηση. Ως Επιτρόπος για τον Προϋπολογισμό, θα αρμόδιος και για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, επίλυση των ε, πολλών προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας χρειαζόμαστε άτομα υψηλής ε, εξειδίκευσης με να μιλούν πολλές γλώσσες και από τα δύο φύλλα και με μια καλή γεωγραφική εκπροσώπηση. Το 2019, στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι στην Αφρία 1,7 ε, ε, μάλλον η Αυστρία αποτελεί 1,7% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 1,5% ε, των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υποεκπροσωπούμενο, ενώ το Βέλγιο, για παράδειγμα, έχει 15% εκπροσώπους στις υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τα συστήματα αυτά για να υπάρξει αποτύπωση και της επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο προσωπικό, στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να δείτε κάποια λύση για να υπάρχει καλύτερη και αναλογικότερη εκπροσώπηση στο προσωπικό. Απάντηση. Είπα ήδη προηγουμένω ότι λίγαν συντόμω θα παρουσιάσω μια στρατηγική για του ανθρώπινου πόρου, HR που θα περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, αλλά και αυτό που αναφέρατε μόλις, ότι υπάρχουν 10 κράτη-μέλη τα οποία υποεκπροσωπούνται. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υψηλές διευθυντικές θέσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς ε, μπορούμε να καταστήσουμε αυτές τις υψηλές θέσεις, τις υψηλότερες θέσεις πιο ελκυστικές. Διαπιστώσαμε για παράδειγμα ότι η Αυστρία, η χώρα μας, κάποια στιγμή σε ό,τι αφορά τι σπουδέ στο κολόγιο τη Μπρουζ, σταμάτησε να τι υποστηρίζετε τι σπουδέ αυτέ. Και ξέρετε ότι στου ε, ειδικού θεωρείται ότι το Κολέγιο τη Ευρώπη αποτελεί ε, το εισιτήριο για να ξεκινήσει κανείς να δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να δούμε πώ θα τα καταστήσουμε πιο ελκυστικά. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν 10 κράτη-μέλη τα οποία δεν εκπροσωπούνται σωστά στι υψηλόβάθμε διευθυντικέ θέσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό καθήκον και θα πρέπει να μα απασχολήσει επισταμένω. Ενδεχομένω, να διοργανώσουμε διαγωνισμούς ε, στοχευμένους ε, σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να εξισορροπηθεί η κατάσταση αυτή σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Τελική ερώτηση. Η Τζάκι Jones από τους σοσιαλιστές. Το καλύτερο έχει μείνει το τελευταίο φανταζόμαι. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Φίλε Ντάγκ, σας ευχαριστώ που επεκταθήκατε για τη ισότητα των φύλων σε σχέση με τη γραπτή απάντηση, χρειαζόταν κάποια διευκρίνηση και για το κράτος δικαίου. Υποσχεθήκατε, υποσχέστε λιγότερα και θέλετε να πετυχαίνετε περισσότερα. Αυτή είναι η αρχή σα. Εγώ θα ήθελα να υπόσχεστε περισσότερα και να δίνετε έτη περισσότερα όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε όλε τι πτυχέ του χαρτοφυλακίου σα. Είχαμε αρκετέ ερωτήσει που αφορούσαν την ισότητα των φύλων. Η προλαλή σα αναφέρθηκε αυτό, η κυρία Πηλία, η Ρουμπιάν και η Βάνα που μου κλέψαν τελικά τις ερωτήσεις μου. Τέλος πάντων, να το θέσω κάπως έτσι το ερώτημά μου. Στην πατρίδα σας είπατε ότι εξετάσατε θετικά τα εργαλεία δημοσιονομικού σχεδιασμού και ποσοστώσεις. Τι άλλο θα εφαρμόσετε σε αυτή την άτυπη ομάδα εργασίας με το Ευρωκοινοβούλιο και με τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Yeah. Ähm, ähm, Αναφερόμουν σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έπρεπε, που είχα αναλάβει εδώ και 12 χρόνια, όταν ανακαλύψαμε ότι ήμουν επιφορτισμένος με τα πανεπιστήμια. Ανακάλυψα τότε ότι οι επιτροπές που ασχολούνται με την ανάθεση εδρών, αν δεν υπήρχε γυναίκα στην Επιτροπή, αυτό είχε αντίκτυπο όσον αφορά τις προδιαγραφές για ενδεχόμενες θέσεις. Ε, προέδρων ή καθηγητών και εδρών. Πρέπει λοιπόν να θεσπίσουμε μια ποσόστοση για να είμαστε σίγουροι ότι οι γυναίκες θα είναι μέλη τέτοιων επιτροπών. Διότι αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στις διάφορες προδιαγραφές στους όρους. Και ανακάλυψα ότι αυτό ήταν που, κάτι που ίσως έπρεπε να θεσπίσουμε και εδώ στις Βρυξέλλες. Αν δεν ισχύει. Αυτό είναι συγκεκριμένο παράδειγμα όπου μπορούμε να επιφέρουμε περαιτέρω βελτιώσεις την ισότητα των φύλων. Άλλο θέμα, Φερρυπίν, υπάρχει κάποια πρωτοβουλία από κάποιους συναδέρφους μου νομίζω, από το Φεβρουάριο τρέχοντος έτους. No woman, no panel λέγεται η πρωτοβουλία. Δεν έχουμε δηλαδή μια επιτροπή, αν δεν υπάρχει η γυναίκα που να συμμετέχει σε αυτήν. Αυτό είναι η φροντίσει όλους μας. Αν προσκληθείτε σε ένα πάνελ να διαπιστώνεται αν υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Θα μπορούσε να είναι και το αντίθετο, να μην έχουμε κανέναν άντρα στο πάνελ, αφού μιλάμε για ισότητα. Αλλά είναι συγκεκριμένα μέτρα αυτά. Τώρα, αν δούμε τα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία πέντε χρόνια. Νομίζω το εντυπωσιακό στοιχείο είναι το εξή. Αν πάρετε το μέσο management, 44% έχουμε γυναίκες εκεί, αύξηση 20% από το 1995. Και τώρα έχουμε πολύ περισσότερες γυναίκες που ξεκινάνε καριέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ότι άντρες, οπότε τελικά όλο και περισσότερες γυναίκες θα είναι στη δίκηση. Για την ώρα όμως κάπως πρέπει να τα σπρώξουμε τα πράγματα. Εν γέννη ο στόχος μας ήταν 40% και τώρα είμαστε 41%. Ευχαριστώ. Τζάκι, την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ για κάποιες από τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Οι ποσοστώσεις είναι μια λύση. Εντό τη άτυπη ομάδα εργασία, παραδείγματο χάρη, θα δεσμευτείτε, να σα βοηθήσω, δεσμευτείτε να βελτιώσετε τι συνθήκε εργασία των Ευρωπαίων ε, δημοσίων υπαλλήλων, των εργαζομένων επί και άλλων υπαλλήλων ούτω ώστε στη στρατηγική σα να έχετε τη διαβούλευση με του κοινωνικού εταίρους, να του λαμβάνετε υπόψη και τι πρώτε 100 μέρε θα δεσμευτείτε να εφαρμόσετε όλε αυτέ τι προτάσει και ελπίζω και περισσότερε. Μπορείτε να πείτε απλώ ένα ναι για να γλιτώνουμε και χρόνο. Τεράστια, τεράστιος πειρασμός αυτός. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω σε 100 μέρες. Συζητήσαμε εξαρτητικά το ποτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, τον προπολογισμό και άλλα τέτοια θέματα. Θέλω να είμαι σοβαρός από την προσωπική μου εμπειρία έχουμε πολλές, πολλούς συμβασιούχους, έξοχους και μετά από 7 χρόνια εκπνέει η σύμβασή τους. Παρά τα ρυθμιστικά και τα μισθολογικά, τη μισθολογική τους θέση εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ συχνά είναι κρίμα να χάνει σε έμπειρον υπάλληλο, γιατί εκείνο ή εκείνη πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από 7 χρόνια είναι ένα θέμα που έχω δική μου εμπειρία και προσπαθώ να αλλάξω τα πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα πώς θα το πετύχουμε αυτό και ποιε θα είναι οι ενδεχόμενε οικονομικές και άλλε συνέπειε, αλλά το γνωρίζω το πρόβλημα που θέσατε. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί. Let me at uh, this... Πρόεδρος, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις τους και για τον υποψήφιο επίτροπο για τις απαντήσεις του. Τώρα θα του δώσω και πάλι το λόγο για την ολοκλήρωση αυτής της ακρόασης. Παρακαλώ να τηρήσετε τα πέντε λεπτά. Έτσι, αυστηρά. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και αν μερικές φορές μακρηγόρησα, ήταν περισσότερο όχι μόνο να δείξω ότι γνωρίζω τα πράγματα, αλλά και από τον ενθουσιασμό μου και την αφοσίωσή μου στα πράγματα. Ίσως μερικές φορές να το ε, παράκανα, αλλά είμαι ιδιαίτερα ενθουσιώδης για αυτό το έργο το οποίο με περιμένει και περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσω. Από τη δική μου την ε, άποψη δεν θεώρησα ότι ήταν ακρόαση ακριβώς αυτό που κάναμε, αλλά μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων που με βοηθάει και εμένα ε, για το έργο μου τους επόμενους μήνες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πάντως ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχω εργαστεί σκληρά και τι να κάνουμε, συγγνώμη που είμαι εδώ ήδη δέκα χρόνια. Θα συνεχίσω πάντως με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον, αφοσιωμένο στο έργο μου σε επαφή με εσάς. Πολλοί από εσά με γνωρίζετε ήδη 10 χρόνια, γιατί κάποιοι από εσά βρίσκεστε εδώ πάνω από 10 χρόνια. Υπάρχει η πολιτική των ε, ανοιχτών θυρών και το τηλεφωνό μου το ξέρετε, μπορείτε να το δώσετε και σε άλλους. Έχω μια πολιτική ανοιχτής προσέγγισης. Είμαι στη διάθεσή σας δηλαδή. Συμμεριζόμαστε πολλές απόψεις και να ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ αφοσιωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για ευρωπαϊκό οικοδόμημα, γιατί έχουμε ήδη προχωρήσει τόσο πολύ. Πρόκειται για ένα θεσμό καταπληκτικό, έναν υπερεθνικό θεσμό. Και μ' αρέσει να εργάζομαι εδώ, να συνεργάζομαι μαζί σας προς το συμφέρον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, προς το συμφέρον των πολιτών μας. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε ότι εργαζόμαστε για τους πολίτες. Μην το ξεχνάμε, να το έχουμε πάντα κατά νου. Ελπίζω να σας έπεισα και να επιβεβαιώσετε τη θέση μου και προσβλέπω στην πενταετή συνεργασία μαζί σας προς το συμφέρον της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. This uh, ends our meeting. Thank Έτσι ολοκληρώνεται η συνεδρίαση αυτή. Οι συντονιστές βέβαια έχουν δουλειά ακόμα, το ξέρουν.